Mes chers collègues, bonjour. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα. Et nous allons... Λοιπόν, συνεχίζουμε τις εργασίες μας. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Μπορούμε να εγκρίνουμε το σχέδιο ημερήσιας διάταξης, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Τα πρακτικά της συνεδρίασης 21ης και 22ης Ιανουαρίου του 2019 Εάν δεν υπάρχουν ενστάσεις μπορούμε να τα εγκρίνουμε. Ανακοινώσει της Προεδρού. Έχετε μεγάλη τύχη διότι δεν έχω να σας πω τίποτα. Ξεκινάμε λοιπόν με το σημείο 4 για το Tourism Task Force αγαπητοί συνάδελφοι. Βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο πολύ σύντομα και θα αρχίσουμε να μιλάμε για χρήματα, για προπολογισμού, για απολογισμούς και για προοπτικές για το μέλλον και ειδικότερα το μέλλον του τουρισμού. Γι' αυτό σήμερα διοργανώνουμε μια τελευταία ανταλλαγή απόψεων εντό τη Ομάδα Εργασία Τουρισμού τη Επιτροπή Μεταφορών με τη φιλοδοξία να συζητήσουμε τα πέντε βασικά επιτεύγματα της ευρωπαϊκής πολιτικής τουρισμού την τελευταία πενταετία και να στραφούμε και λίγο προς το μέλλον, να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Ο τουρισμός ε, αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της ευρωπαϊκής πολιτικής. Μην ξεχνάτε ένα συνέδριο υψηλού επίπεδου το 2017 για τον τουρισμό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την ευκαιρία της Διεθνούς ημέρας τουρισμού. Επιπλέον τον Νοέμβριο του 2018 στην Ολομέλεια ζητήθηκε να υπάρχει μια δημοσιονομική γραμμή για τον τουρισμό στο επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η δική μας Επιτροπή εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση και σήμερα θα ήθελα να καλωσορίσω τους εξής προσκεκλημένους, την κυρία Άννα Αθανασοπούλου, Ευχαριστούμε που βρίσκεστε μαζί μας. Είστε επικεφαλής του Τμήματος Τουρισμού ε, αναδιόμενων και Δημιουργικών Βιομηχανιών στην DG Grow, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστούμε που είχατε την καλοσύνη να έρθετε να μας επισκεφτείτε στην Επιτροπή μας. Μετά έχουμε τον κύριο Εντουάρδο Σανταντέρ. Καλώς ορίσατε στην Επιτροπή μας. Είστε ο εκτελεστικός διευθυντής της European Travel Commission, ETC. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Οι προσκεκλημένοι μα θα μας κάνουν ε, σύντομες παρουσιάσεις ε, για το πολύ σημαντικό αυτό θέμα για την Επιτροπή μας, τον τουρισμό. Αγαπητοί ομιλητέ, ήθελα να σας πω ότι έχετε 7 λεπτά στη διαθέσή σα ο καθένα. έχουμε περιορισμένο χρόνο για να μας ε, κάνετε τις παρουσιάσει σα και μετά θα δώσουμε το λόγο στους βουλευτές οι οποίοι θα σας κάνουν και ερωτήσει. Δίνω όμως πρώτα το λόγο στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής μας και Πρόεδρο της Ομάδας Εργασίας του Τουρισμού, τον κύριο Ούρικε. Είστε εδώ για να μας παρουσιάσετε με πιο συγκεκριμένο τρόπο όλες τις στοιχείες του τουρισμού τα τελευταία δεκαετία. Κύριε Χέλγε, έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητή Άννα, αγαπητέ καλώς ορίζω τους πάντες και εσάς και τους προσκεκλημένους και τους επαγγελματικούς οργανισμούς, όλους ενδιαφερομένους που ήρθαν εδώ πέρα και μας θυμούν με την παρουσία τους σήμερα. Προετοιμάζοντας την τελευταία μας ε, συνεδρίαση της Task Force, έριξα μια ματιά στο παρελθόν για να δω τι έχει γίνει την τελευταία πενταετία. Και αισθάνθηκα χαρούμενος κάνοντας έναν απολογισμό των όλων έχουμε, όσων έχουμε επιτύχει εμείς εδώ ε, στο, για τον τουρισμό στην Επιτροπή μας και ως Κοινοβούλιο. Ε, δύο είναι τα βασικά κεφάλαια. Το πρώτο η Επιτροπή ΤΡΑΝ συνέβαλε στις νομοθετικές εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, για συμμετοχή στις τακτικές, για να το πω έτσι, βουλευτικές δραστηριότητες. Ε, πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι ο τουρισμός δεν είναι θέμα για το οποίο συνεδριάζουμε κάθε εβδομάδα για να μιλήσουμε για νομοθετικά θέματα. Στην τρέχουσα θητεία όμως ε, πολλές φορές ε, έχουμε εκφράσει τις απόψεις μας είτε πρόκειται για τη δεσμή μέτρων για τις θεωρήσεις ε, είτε πρόκειται για άλλες πτυχές όπως ελεία όπως η συνεργατική οικονομία Η Επιτροπή μας ε, και οι αγαπητοί μου συνάδελφοι λοιπόν έχουν συμβάλει με το δικό τους τρόπο και τις δραστηριότητες τους σε πολλά διαφορετικά θέματα. Το σημαντικό τροπόνημα ήταν ε, η σχετική έκθεση για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο τουρισμός. Και ευχαριστώ και τους συναδέλφους για τις προσπάθειές τους. Αν και ξέρετε, το πραγματικό αποτέλεσμα δεν είναι το αποτέλεσμα εδώ το, ως κοινοβουλευτικό έργο. Το αποτέλεσμα, το πραγματικό είναι το αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων μας, ε, lobbying ουσιαστικά. Τι έχουμε κάνει λοιπόν την τελευταία πενταετία. Είχαμε πέντε υπουργικές ε, ε, συναντήσεις, ε, πέντε άτυπα συμβούλια, τα οποία διοργάνωσε η Προεδρία του Συμβουλίου η και όπου η Επιτροπή Τραν είχε στείλει επαρκή αντιπροσώπευση. Πολλές φορές υποδεχθήκαμε εδώ τον εκάστοτε Επίτροπο Τουρισμού και κάτι καινούριο κάτι που δεν είχε επαναληφθεί στο παρελθόν. Στήσαμε μια στρατηγική συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα της Παγκόσμιας Τουρισμού, του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, ε, με τους εκπροσώπους του WTC, με πρωτοβουλία δηλαδή της Επιτροπής μας, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου σύναψε συμφωνίες συμφωνίες που αποδεικνύουν απτά τις ευθύνες που έχουμε αναλάβει στον τομέα του τουρισμού και που έτυχαν ιδιαίτερα σε εκτίμηση στον κλάδο. Εμβαθύναμε τις επαφές μας με την Επιτροπή των Περιφερειών σε θέματα τουριστικά. Διοργανώσαμε πολλές και διάφορες εκδηλώσεις και δράσεις στα οποία συμμετείχαν ε, οι συναδελφοί μας από το Κοινοβούλιο και εκπρόσωποι της Επιτροπής των Περιφερειών. Επίσης είχαμε την ευκαιρία να εκφέρουμε απόψεις σε, για διάφορες, ε, σε διάφορες εκθέσεις της Επιτροπής των Περιφερειών. 11 εκατομμύρια ευρώ αφιερώθηκαν, δόθηκαν μάλλον σε ε, πιλωτικά έργα και σε άλλες πρωτοβουλίες. Πρωτοβουλίες σχετικές ε, με τον τουρισμό. Ξεκίνησαν και διάφορα προγράμματα μετά από πρωτοβουλίες ε, των συναδέλφων μας εδώ στην Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με διαβεβαίωσε ε, ότι ουδέποτε στις παλιότερες θητείες δεν είχε διασφαλιστεί τέτοιο ποσό για τον τουρισμό ε, και για πιλωτικά έργα στον κλάδο αυτών. Ε, η κυρία Πρόεδρος λοιπόν ε, αντιλήφθηκε πόσο μεγάλη ήταν η επιτυχία μας και έτσι το περασμένο Οκτώβριο καταφέραμε να διασφαλίσουμε μια δημοσιονομική γραμμή, ένα κονδύλιο δικό για τον τουρισμό. Το Κοινοβούλιο οργάνωσε μια μεγάλη δράση με τη συμμετοχή του Πρόεδρου του Κοινοβουλίου πρόκειται για την ημέρα τουρισμού. Για τη διάσκεψη υψηλού επίπεδου για τον τουρισμό με την ευκαιρία της ε, Διεθνούς ημέρας τουρισμού. Εκεί ξεκίνησε μια ολόκληρη σεζόν τουριστική, για να το πούμε έτσι, εδώ στο Κοινοβούλιο. Για να σας δώσω και κάποια τελευταία νούμερα που συμπληρώνουν την εικόνα, ήθελα να σας υπογραμμίσω ότι αυτό που είναι σημαντικότερο για μένα είναι οι καθημερινές επαφές που δημιουργήθηκαν και που συνεχίζονται με τις επαγγελματικές οργανώσεις στον τομέα του τουρισμού. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο Γενικός Γραμματέας του ETC και η εκπρόσωπος εδώ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, συμμετέχουν εδώ σε αυτή τη συνεδρίαση σήμερα. Υπάρχει ο κύριος Ανταμποτό που είναι παρόν εδώ και άλλοι επαγγελματίε του κλάδου του τουρισμού. Έχουμε θέσει ως στόχο να υιοθέσουμε κάποιο είδους ε, κοινό μανιφέστο. Το ε, κοινό για όλους τους οργανισμούς ε, και τα θεσμικά όργανα. Αυτό θα είναι το σημαντικό αποτέλεσμα που θα προκύψει από αυτή μας τη θητεία, από αυτόν τον κύκλο. Το γεγονός λοιπόν ότι καταφέραμε να εκπονήσουμε αυτό το έγγραφο όλοι μαζί είναι από τις σημαντικότερες επιτυχίες. Μεγαλύτερη επιτυχία από οποιοδήποτε νομοθέτημα. Το μήνυμα που προσπαθώ να δώσω δεν είναι ότι ήταν σημαντικό το ότι έχουμε στα χέρια μας ένα χαρτί αλλά το γεγονός ότι Καθημερινά είχαμε επαφές ε, με, τον διαφόρων, τους εκπροσώπους των διαφορών οργανισμών. Πρέπει λοιπόν να συνεχιστεί το ίδιο και στο μέλλον, να συνεχιστεί η συνεργασία με τους επαγγελματίες του κλάδου. Εγώ σε 35 διαφορετικές εκδηλώσεις και δράσεις εκπροσώπησα την Επιτροπή Τραν εκτός των Βρυξελών Οργανώσαμε μάλιστα και 200 εκδηλώσεις εδώ στις Βρυξέλλες. Ευχαριστώ λοιπόν για όλη αυτή την κοινή προσπάθεια. Ευχαριστώ όλους σας. Και σας υπενθυμίζω να μην ξεχνάμε να ευχαριστήσουμε και τον UNWTO και τον κύριο Γενικό Γραμματέα. Έχω πρόθεση να συνεχίσω το ε, νομοθετικό μου έργο και το κοινοβουλευτικό μου έργο και μετά τις 25 Μαΐου και να συνεχίσουμε και το κοινό μας έργο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πλέον όλοι ξέρουν ότι είστε υποψήφιο. Και τώρα θα ακούσουμε τους εμπειρογνώμονές μας. Η κυρία Θανασοπούλου έχει το λόγο για 7 λεπτά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αξιότιμοι φίλοι. Λόγω τη οζόντια φύση του, μια σειρά από πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση συνδέονται με τον τουρισμό. Ενιαία αγορά, ψηφιακή ενιαία αγορά, βιομηχανική πολιτική, προστασία καταναλωτή, μεταφορέ, ενέργεια, περιφερειακή πολιτική, δεξιότητε και εκπαίδευση, φορολόγηση, πολιτική θεωρήσεων για να πω τα πιο σημαντικά. Γι' αυτό τον λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να ευθυγραμμίσει τα συμφέροντα ε, τον, τον, του τομέα του τουρισμού σε διάφορε πολιτικέ μα και να υπάρχει συμπληρωματικότητα μεταξύ των μέτρων στηρίξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τον τουρισμό αποτελεί μέρο μια σφαιρική προσέγγιση. Τα τελευταία πέντε χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποβάλει μια σειρά από προτάσει που σχετίζονται με τον τουρισμό και η Επιτροπή μας έχει ασχοληθεί με αυτό. Επίσης προτείναμε να κινητοποιήσουμε διάφορα χρήματα, διάφορα ταμεία που σχετίζονται με, το, τον τουρισμό. Στα πλαίσια του, του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης πάνω από 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ ε, έχουν διατεθεί για τον τουρισμό έως το 2020. Επιπλέον, πέρα από αυτές τις οριζόντιες δράσεις, δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναπτύξει εστιασμένες δράσεις που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό. Και θα ήθελα σήμερα να επικεντρωθώ σε αυτό το σκέλος, στην πολιτική τουρισμού ε, ένας τομέας όπου είναι περιορισμένε οι αρμοδιότητε της Ένωσης για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων τουρισμού και να αναπτύξουμε δράσεις οι οποίες είναι συμπληρωματικές αυτές των κρατών μελών. Το σχετικό κονδύλιο ε, προέρχεται από το COSME. Μιλάμε για 42 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2014-2019. Για την ίδια περίοδο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εφαρμόσει μια σειρά από πιλωτικά προγράμματα που σχετίζονται με τον τουρισμό για ένα ποσό 11,5 εκατομμυρίων ευρώ. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτή την Επιτροπή ιδιαίτερως που υπέβαλε τις προτάσεις αυτές. Χάρη στην ενεργή συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αυτής της Επιτροπής έχουμε δημιουργήσει ε, μια έντονη και επικοδομητική συνεργασία που έχει φέρει αποτελέσματα. Πρώτα απ' όλα ε, έχουμε μια κοινή σε ό,τι αφορά τι βασικέ πολιτικέ προτεραιότητε στον τομέα του τουρισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμεί επικεντρωνόμαστε σε αυτέ τι ε, τομέ προτεραιότητα, ε, Υπάρχει ένα ευρύτερο βέβαια πολιτικό πλαίσιο που καθορίζει η, ε, η ανακοίνωση του 2010 ε, για τον τουρισμό, το κείμενο του 2017 και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προώθηση του τουρισμού στην Ευρώπη του 2015. Αυτέ οι πέντε, προτε... πέντε προ... είναι οι εξή. Πρώτα απ' όλα προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις ε, συνθήκες και το πλαίσιο, το ρυθμιστικό πλαίσιο και να ενισχύσουμε τις έξυπνε επενδύσεις. Δεύτερον, ε, δίνουμε έμφαση στον έξυπνο τουρισμό, και στην καινοτομία του τουρισμού, να συνοδεύσουμε ε, τον, την τουριστική βιομηχανία στην ψηφιακή εποχή, καθώς και την sharing economy. Τρίτον, Βιώσιμο και υπεύθυνο τουρισμό. Υποστηρίζουμε τη βιωσιμότητα του τουρισμού, αποτελεσματική χρήση ενέργεια, κυκλική οικονομία, τουριστικέ ροέ, τουριστικές ροές και διαφοροποίηση των τουριστικών προϊόντων. Τέταρτον, επικεντρωνόμαστε στην ανθεκτικότητα του ε, εργατικού δυναμικού του τουρισμού, να βελτιωθεί οι δεξιότητέ του και η ποιότητα τη εργασία του. Και πέμπτον, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τι προκλήσει του παγκόσμιου ανταγωνισμού, υποστηρίζοντα την διεθνοποίηση των τουριστικών επιχειρήσεων και προωθώντας την Ευρώπη ως τουριστικό προορισμό. Στα υπόλοιπα λεπτά θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια παραδείγματα στα πλαίσια της κάθε προτεραιότητα για να σας δείξω ποιο είναι το εύρο των ε, πρωτοβουλίων που έχουμε πάρει τα τελευταία πέντε χρόνια. Για την πρώτη προτεραιότητα πρώτα, δηλαδή ε, το γενικότερο πλαίσιο και τις προϋποθέσεις. Η προσέγγιση ή μάλλον η πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι κρίσιμη εδώ, γι' αυτό έχουμε ετοιμάσει έναν λεπτομερή οδηγό για τη χρηματοδότηση του τουρισμού που είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες της Ένωσης για να βοηθήσουμε ε, τους εμπλεκόμενους φορείς στον τουρισμό να εξετάσουν τις διάφορες πηγές ε, χρηματοδότησης που είναι διαθέσιμες στον τομέα του τουρισμού. Στα πλαίσια του προγράμματος COSME υποστηρίξαμε πάνω από 100 ε, διεθνής ε, συμπράξεις όπου συμμετέχουν πάνω από 150 ε, μικρές επιχειρήσεις και 200 ευλεκόμενοι φορείς από 31 ευρωπαϊκές χώρες. Καινοτόμες προ, προτάσεις, βιώσιμες, πολιτιστικές, ε, σε ό,τι αφορά τον παράκτιο τουρισμό μεταξύ άλλων. Στα πλαίσια της ε, πλατφόρμας για την έξυπνη ε, ψηφιοποίηση. Αυτή τη στιγμή συνεργάζονται 18 επιχειρήσει μαζί μα για να μπορέσουν να βελτιωθούν δυνατότητε καινοτομία και να αναπτύξουμε προγράμματα επενδύσεων για την ψηφιοποίηση και τη χρήση των big data, καθώ και το θέμα τη ασφάλεια στον τομέα του τουρισμού. Σε ό,τι αφορά τώρα τη δεύτερη προτεραιότητα, τον έξυπνο τουρισμό, καινοτομία, ψηφιακή ε, μεταβή, με, μετάβαση, ψηφιακή οικονομία. Να δώσω κάποια παραδείγματα και εδώ. Πρώτα απ' όλα χρηματοδοτούμε το, για πρώτη φορά ένα διεθνές ε, δίκτυο incubator. Συμμετέχουν 10 εταιρεία από 9 κρατημέλη που υποστηρίζουν ε, την βελτίωση και την ε, ενίσχυση των startup στον τομέα του τουρισμού. Το 2015 δημιουργήσαμε και το δίκτυο ψηφιακού τουρισμού για να προσθεθεί ο διάλογο ευρωπαϊκό επίπεδο για τι προκλήσεις και τι ευκαιρίε τη ψηφιοποίηση στον τουρισμό. Δύο ακόμα συνεδριάσεις αυτού του δικτύου προβλέπονται φέτος. Επίσης, έχουμε εστιασμένη υποστήριξη για δημιουργία δυνατοτήτων σε ό,τι αφορά τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, τι τουριστικέ, μέσω κάποιων webinars που οργανώσαμε. Αυτό που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι ότι πάνω από 120.000 ε, άνθρωποι, επιχειρηματίε του τουρισμού, παρακολούθησαν αυτά τα τα webinars και είχαμε και τοπικά σεμινάρια όμως που οργανώθηκαν σε πέντε κράτη-μέλη. Επίσης αναλάβαμε δράσεις σε ό,τι αφορά τη συνεταιριστική οικονομία, σε ό,τι αφορά το μακροπρόθεσμο, τον βραχυπρόθεσμο τομέα, τον τομέα της βραχυπρόθεσμης ενοικίασης. Οργανώσαμε εργαστήρια για να δούμε πώς θα εφαρμοστεί η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και να καθορίσουμε κάποιε βέλτιστε πρακτικέ ό,τι αφορά τη ρυθμιστική προσέγγιση. Γι' αυτό οδήγησε σε κάποιε αρχέ για του εφαρμοστέου κανόνε σε ευρωπαϊκό επίπεδο που παρουσιάστηκαν τον περασμένο Οκτώβρη στην διάσκεψη ψηλού επίπεδου που οργανώθηκε στι Βρυξέλλε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή συνεχίζει το διάλογο με του εμπλεκόμενου φορεί για να παρακολουθήσει την εξέλιξη τη ε, συνεταιριστική οικονομία στον τομέα ε, τη ε, στέγαση. Ε, πάντα στον έξυπνο τουρισμό ε, επειδή όταν μιλάμε για ε, έξυπνο τουρισμό ε, έχουμε αποφασίσει οι πρόσφατες δράσεις της Ένωσης οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, τουρισμού να ενισχυθούν. Το Ελσίνκι και η Λιόν λοιπόν είναι οι πρώτες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έξυπνου τουρισμού του 2019 επελέγησαν από 38 πόλεις από 19 κράτη-μέλη. Ε, έχει ξεκινήσει ο διαγωνισμό για το 2020 από πέρυσι, από την προηγούμενη εβδομάδα, συγγνώμη, έω τι 20 Μαου. Ελπίζουμε μέσω τη πρωτοβουλία αυτή να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα ευρωπαϊκών πόλεων που είναι διατεθειμένε να αλλάξουν εμπειρίε για να αναπτύξουν τον έξυπνο τουρισμό και να μάθουν οι μένα από του δε. Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ στην τρίτη προτεραιότητα. Βιώσιμο και υπεύθυνο τουρισμό. Είναι αλήθεια ότι η βιωσιμότητα αφορά τον τουρισμό ποικιλοτρόπω, περιβαλλοντικά, οικονομικά, κοινωνικό, κοινωνικά. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε να ενισχύσουμε την ε, στήριξη στα πλαίσια του προγράμματο Κόσμου για πρώτη φορά φέτο, κινητοποιώντα 5 εκατομμύρια ευρώ ε, για να βρεθούν καινοτόμε λύσει και δημιουργία αναρωτήτων στον βιώσιμο τουρισμό αυτή η υποστήριξη έχει να συμπληρώσει τις εργασίες μας για την πρόθεση του, του, του, του βιώσιμου τουρισμού μέσω προγράμματος όπως το ΕΘΙΣ, που είναι ένα εθελοντικό πρόγραμμα δικτών που είναι στη διάθεση των πλουστικών προορισμών ή μέσω του Eden, ε, το, που αφορά το δίκτυο αριστείας που προωθεί λιγότερο γνωστούς τουριστικούς προορισμούς. Επίσης, ανθεκτικότητα των ε, εργαζομένων, η ανάπτυξη δεξιοτήτων. Προσπαθήσαμε εδώ να δούμε ποια είναι τα, ποια είναι τα κενά σε δεξιοτήτων στον τουρισμό. Το χαρτογραφήσαμε και το 2017 βάσει αυτού ξεκινήσαμε ένα blueprint για τη συνεργασία δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού. Έτσι ώστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να μπορέσουμε να προβλέψουμε αυτέ τι δεξιότητε και να τι αναπτύξουμε. Ελπίζουμε το αποτέλεσμα αυτή τη εργασία να φανεί σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο μετά το 2020 όταν θα ολοκληρωθεί το project αυτό. Θα ήθελα τώρα να φτάσω στην τελευταία προτεραιότητα, διεθνοποίηση και παγκόσμιος ανταγωνισμός. Είναι αλήθεια ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί 40% του, του, της αγοράς ε, του τουρισμού, όμως το μερίδιό μας μειώνεται, διότι υπάρχει παγκόσμιος ανταγωνισμός. Γι' αυτό λοιπόν επικεντρωνόμαστε στο να προωθήσουμε τον προορισμό Ευρώπη στις αγορές ε, τις μακροπρόθεσμες ε, και ιδιαίτερα να προωθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για την προώθηση χρησιμοποιούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδίων που ειδικεύεται σε αυτό. 12,7 εκατομμύρια, εκατομμύρια έχουν διατεθεί για την περίοδο 2014-2021. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα κοινό, μια κοινή πλατφόρμα προώθησης, ένα νέο εργαλείο συνεργασίας που με εκστρατείες online, offline, με ποικίλου τρόπου ε, να δείξουμε ότι υπάρχει μεγάλη προσφορά τουριστική. Η πρόθεση όμω δεν αρκεί εάν δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε δυνατότητε για τι επιχειρήσει να έχουν πρόσβαση σε νέε αγορέ. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε υποστηρίξει τη διεθνοποίηση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων τουρισμού, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με έναν προπολογισμό 3,1 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω των, του οποίου οργανώσαμε ε, κάποιες εκδηλώσεις matchmaking το 2018 και το 2019. Το 2019 πιο συγκεκριμένα με, τον, ε, με την χρονιά τουρισμού της Κίνα, Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας μπορούσαμε να προωθήσουμε το θέμα αυτό της διεθνοποίησης και να το ε, εφαρμόσουμε. Το πρώτο, αποτέλεσμα, το πρώτο αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών είναι αρκετά θετικά. Ε, διαπιστώνουμε 7,9% αύξηση αφήξεων από την Κίνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τους τελευταίους τέσσερις μήνες του 2019 και υπάρχει μια σημαντική αύξηση κρατήσεων για το πρώτο, τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2019. Ίσως η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή Ταξιδίων να μπει σε λεπτομέρειες από αυτού. Σε ό,τι αφορά τώρα τα αποτελέσματα του, της, του έτους Ένωση τη Κίνα από προβάσει επιχειρήσεων για πρώτη φορά φέραμε κοντά περίπου χίλιε ε, ευρωπαϊκές 850 κινέζικες επιχειρήσει, ε, ε, σε μεγάλα σαλόνια τουρισμού και ταξιδίων και, και πάνω από 450 πρωτοβουλίες έλαβαν χώρα σε εθνικό, τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και σε διεθνές επίπεδο. Αυτό δεν, δεν σταματάει. Το 2019 θα συνεχίσουμε ε, τη συνεργασία με τις κοινωνικές αρχέ για να ενισχύσουμε τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, τουρισμού και να υπάρξει αμοιβαία κατανόηση. Και φτάνω τώρα ε, στο μέλλον και θα κλείσω με το μέλλον. Καθώ εξετάζουμε λοιπόν το μέλλον, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με βάση τι προτεραιότητε που παρουσιάσαμε σήμερα. Γιατί? Διότι θα συνεχίσουμε το mainstreaming, να κάνουμε mainstreaming του τουρισμού στι ευρωπαϊκές Πολιτικέ, ε, παγκόσμιος ανταγωνισμό, βιωσιμότητα, αυτά είναι οριζόντια ζητήματα. Ε, αυτή η οριζόντια σφαιρική προσέγγιση αποτυπώνεται άλλωστε στην πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το επόμενο πολιτές μεσονομικό πλαίσιο, ε, όπου ελπίζουμε ότι θα έχουμε πλήρη και σφαιρική στηρίξη σε διάφορους τομείς όπως τον τομέα της συνοχής, ε, InvestEU, Horizon Europe, ε, το πρόγραμμα Νέα Αγορά και το πρόγραμμα Creative Europe. Βεβαίως οι διαπραγματεύσει για το πάνω πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο είναι εξελίξη. Ελπίζουμε το αποτέλεσμά τους ε, να εξασφαλίσει την κατάλληλη χρηματοδότηση του τουρισμού για το επόμενο πολιτή δημοσιονομικό πλαίσιο και από κοινού με του συναδέλφου ε, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εμεί ε, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την, ε, τον ευρωπαϊκό τουρισμό και τι μικρομεσαίε επιχειρήσει στο μέλλον. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη που σα διέκοψα προ στιγμή. Είναι σημαντικό για μα το θέμα, αλλά ε, θα ήθελα ο Εντουάρντο που θα πάρει το λόγο τώρα να μιλήσει όντω 7 λεπτά. Θα σου φτάσουν, Εντουάρντο. Παρακαλώ. Έχεις το λόγο, Εντουάρντο Σανταντέρ. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πολύ Ιστβάνε που με καλέσατε σήμερα εδώ και αποδέχτηκα φυσικά αυτή την ε, πρόσκληση όχι μόνο εκ μέρους ε, ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του ταξιδιωτικού τομέα αλλά και εκ μέρους του Μανιφέστο. Έτσι λοιπόν εγώ Δημής δηλαδή μου βρίσκομαι σήμερα εδώ αλλά δεν εκπροσωπώ μόνο ε, το μανιφέστο αλλά και την επιτροπή και πραγματικά είναι η τιμή μου που ε, τους εκπροσωπώ σήμερα εδώ. Γιατί λοιπόν χρειαζόμαστε ένα μανιφέστο. Καταρχήν να σας υπενθυμίσω ε, τους λόγους για τους οποίους ε, ξεκινήσαμε αυτή την πρωτοβουλία και με την ε, ισχυρότατη υποστήριξη από την πλευρά πολλών μελών εδώ του Ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου και ειδικώς ε, του, του Ιστβάν Ουλιέ. Καταρχήν επειδή ο κλάδος μας είναι η πάρα πολύ κατακαιρματισμένος και αυτό θεωρείται βέβαια ως ένα μειονέκτημα από την πλευρά του, του κλάδου μας. Δηλαδή μας λένε συχνά τα θεσμικά όργανα ότι ε, είσαστε πολλοί από εσά και ζητάτε τα ίδια πράγματα. Πώς μπορούμε λοιπόν να τα αποκριθούμε σε όλα σας τα αιτήματα. Άρα θα πρέπει λοιπόν να μιλάμε με την ίδια φωνή. Και από εκεί και μετά χρειαζόμασταν και κοινού στόχους γιατί τα μεγάλα επιτεύγματα είναι πραγματικά τα συλλογικά και γι' αυτό ακριβώς το λόγο ε, και με αυτό το σκεπτικό καταφέραμε να δείξουμε ένα κοινό μέτωπο, να μιλήσουμε με την ίδια φωνή αλλά να σας δείξω το, καταρχήν το γιατί είναι ε, πολύ σημαντικός αυτός ο κλάδος. Βέβαια γνωρίζετε όλη την σημασία εδώ μέσα σε αυτή την αίθουσα του τουρισμού, αλλά ποτέ δεν κουράζομαι να επαναλαμβάνω ε, τα ωφέλη ε, του κλάδου, γιατί πραγματικά είναι τεράστια για τους πολίτες μας, αλλά και για την οικονομία μας, αλλά και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την προώθηση της ανάπτυξης που τόσο χρειαζόμαστε. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε παρά να επαναλαμβάνουμε αυτήν τη σημασία του ε, τομέα τόσο εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε αυτήν εδώ την Επιτροπή αλλά και εκτός ε, του Κοινοβουλίου σε όποιους ε, ενδιαφέρονται γιατί για κάποιους ο τουρισμός αντιστοιχεί μόνο στο να πηγαίνουν σε μια ωραία παραλία ή σε ένα ωραίο τουριστικό μέρος. Πάντω, εσκεμένα δώσαμε την ονομασία σε αυτή την πρωτοβουλία τουρισμό για την ανάπτυξη και τι θέσει εργασία, γιατί ακριβώ γνωρίζαμε και ότι αυτέ είναι κύριε προτεραιότητε τη Επιτροπή ε, του κ. Γιόνκερ και θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να ευθυγραμμίσουμε λοιπόν τι δικέ μα προτεραιότητε με τι προτεραιότητε τη Επιτροπή Γιόνκερ. Οι δικέ μα ε, λοιπόν ε, προτεραιότητες που θέτουμε εδώ παραμένουν πάρα πολύ σημαντικέ, δηλαδή η ανταγωνιστικότητα, η ψηφιοποίηση, η καλή διακυβέρνηση, η προώθηση τη Ευρώπη ω τουριστικού προορισμού, η βιωσιμότητα, η βελτίωση των δεξιοτήτων, η διασυνδεσιμότητα. Όλα αυτά λοιπόν τα συζητούμε ξανά και ξανά εδώ στην Ευρώπη και ίσω εντάξει κάποια από αυτά ακόμα να μην τα συζητάμε στο βαθμό που πρέπει σε ό,τι αφορά τον ε, τουρισμό, αλλά ε, νομίζω ότι θα φτάσουμε εκεί. Ε, όταν ε, ξεκινήσει αυτή την πρωτοβουλία θα ήθελα να ευχαριστήσω εδώ τον ε, συνάδελφο από την ε, Ομοσπονδία European Cycle Federation ε, που είχε μαζί μου την ιδέα του να ξεκινήσουμε αυτή την πρωτοβουλία και σήμερα έχουμε 45 συμμετέχουσες οργανώσεις οι οποίες προέρχονται και από τον τομέα των χερσαίων μεταφορών, των θαλάσσιων, των αεροπορικών μεταφορών, των, της εστίασης, των ξενοδοχείων, των ταξιδιωτικών πρακτόρων, τουριστικών αξιοθέατων και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν μιλάμε όλοι με μια κοινή φωνή και ε, και είμαστε εδώ για να σας ακούσουμε αλλά και για να δώσουμε καθοδήγηση. Ε, είμαστε από τη μία πλευρά τώρα μία άτυπη ομάδα αλλά δημιουργήσαμε μία επίσημα θέλετε δομή ε, και Παρότι λοιπόν δεν υπάρχει επίσημη συμμετοχή μελών, έχουμε μια δομή η οποία μας επιτρέπει να λειτουργούμε αποτελεσματικά. Εγώ είμαι λοιπόν ο πρόεδρος και έχω δύο αντιπροέδρους και έχω και εδώ και τον συνάδελφο Γιουλέν Κούλιτσα, ο οποίος προσωπεί τη γραμματεία και διοργανώνει δηλαδή τα πράγματα παρασκηνιακά αν θέλετε και εδώ στις ε, Βρυξέλλες. Η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα ε, του τουρισμού, European Travel Commission, με τα τιμή έχει αναλάβει λοιπόν την προεδρία αυτή τη άτυπη ομάδα και θα την κρατήσει στο βαθμό που αυτό είναι επιθυμητό, γιατί πραγματικά είναι σημαντικό να δείξουμε και συνέχεια στο πλαίσιο τη τρέχουσα βουλευτική ε, περίοδου. Να σα δώσω τώρα κάποιε σύντομε πληροφορίε ω προ τα όσα έχουμε κάνει τώρα τελευταία. Άρα λοιπόν από τότε που ε, δημιουργηθήκαμε το 2015 Είχαμε καταρχήν τη φάση, αν θέλετε, του ευαγγελισμού εντό εισαγωγικών. Δηλαδή, τι προσπαθήσαμε να κάνουμε. Αρχίσαμε να συναντιόμαστε όχι μόνο με τον αρμόδιο επίτροπο, αλλά όπω λάβαμε και τι σχετικέ ε, ε, συμβουλέ, ε, ήρθαμε και σε επαφή και με τους αρμόδιους από το τομέα του πολιτισμού και τον Επίτροπο Τιμπον και πράγματι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η ενοποίηση αν θέλετε των πολιτικών γιατί για παράδειγμα ένα μουσείο χωρίς ακριβώς να ε, αποτελεί και πόλο έλξη σε τουριστικό επίπεδο είναι ένα άδειο μουσείο. Επίσης είχαμε και κάποιες ακροάσεις και στο πλαίσιο της Task Force για τον τουρισμό ε, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συνεργασία με την δική σας ε, την Επιτροπή φυσικά το 2017 ε, αποστήλαμε μια ανοιχτή επιστολή στον πρόεδρο Γιούντερ από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή των Περιφερειών για το θέμα του τουρισμού, στην οποία όμως από αποστολή δεν λάβαμε ποτέ απάντηση. παρόδο. Ε, τώρα, τι κάναμε ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση το 2018, δηλαδή πιο πρόσφατα. Είχαμε καταρχήν ω ένα μεγάλο επίτευγμα ε, τη θέση μα σε ό,τι αφορά τον εξυγχρονισμό τη πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ό,τι αφορά τι θεωρήσει ε, βραχία περίοδου, μικρή περίοδου. Γιατί βέβαια και μια τέτοια περισσότερη ευελιξία σε σχέση με αυτέ τι πολιτικέ έχουν σημαντικό ρόλο για τον κλάδο του τουρισμού. Άρα λοιπόν το εκείνο που, είναι, που θα πρέπει να αποφύγουμε είναι όχι να μειωθεί το μερίδιο της αγοράς της Ευρώπης στον κλάδο ε, του τουρισμού, αλλά να μειωθεί η ανταγωνιστικότητά μας και αυτό είναι που συμβαίνει. Επίσης ε, ζητήσαμε να υπάρξει στο επόμενο ε, πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021 έως 2027 η περισσότερα κονδύλια και γραμμή του υπολογισμού συγκεκριμένα για τον τουρισμό. Ε, και βέβαια όλα αυτά ε, τα οποία καταφέραμε δεν τα επιτύχαμε μόνοι μας ε, και είχαμε πάρα πολλούς συναδέλφους που μας υποστήριξαν. Όχι η κυρία Μοντέρο, η κυρία Ντελμόντ, η κυρία Τοπαρδέλα και άλλοι, άλλα μέλη εδώ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν ασκήσει αντίστοιχες πιέσεις μαζί μας. Τώρα, άλλα επιτεύγματα τα οποία σημάδεψαν τα όσα κάναμε κατά τα τελευταία χρόνια είναι ότι ε, προωθήσαμε την πρόταση που έγινε ούτως ώστε να έχουμε απλούστερες και πιο ευέλικτους κανόνες σε ό,τι αφορά τις θεωρήσεις αλλά και την ε, αύξηση των κονδυλίων για τον τουρισμό κατά 300 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό λοιπόν αποτελεί ε, αποτέλεσμα των προσπαθειών που κάναμε από κοινού και εδώ με τα μέλη της Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και βέβαια ήταν πολύ σημαντική και η υποστήριξη από τα θεσμικά όργανα. Και ευχαριστώ θερμά την κυρία Θανασοπούλου για την ε, πραγματικά πολύτιμη ε, βοήθεια που μας ε, παρήχε, αλλά ευχαριστώ την κυρία Κουράτσα. Και θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω τον κύριο Ορτούν, ο οποίος πραγματικά αποτέλεσε έναν από τους πατέρες, αν θέλετε, αυτού του μανιφέστο και πραγματικά τον ευχαριστούμε. Και φυσικά συνέβαλαν όλοι εδώ οι βουλευτές ε, αλλά και ε, ο πρόεδρος Σταγιάννη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν πάντοτε διατεθειμένος να υποστηρίξει και επέδειξε μεγάλη υποστήριξη απέναντι στον ε, τουρισμό ασχέτως πολιτικής ομάδας, ασχέτως κατεύθυνσης και μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα του διαβιβάστηκε ένα έγγραφο κληρονομιάς, αν θέλετε, ένα legacy paper ούτως ώστε να δώσουμε τη δική μας άποψη ως το πιο ποιο θα πρέπει να είναι το μέλος του τουρισμού και ότι θα πρέπει να αυξηθεί ο, ο προϋπολογισμός ε, ε, για τον τουρισμό στο επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ε, σε ό,τι αφορά αυτή την ξεχωριστή γραμμή του προϋπολογισμού στον στο μέλλον θεωρούμε πως θα συμβάλλει με αυτόν τον τρόπο να παραμείνουμε πιστοί στην ατζέντα που έχουμε θέσει και απέναντι σε όσους μας υποστηρίζουν και ελπίζουμε ε, πως ε, η Επιτροπή Τραν και στο πλαίσιο του επόμενου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα συνεχίσει να μας υποστηρίζει και βέβαια ε, εύχομαι καλή τύχη σε όλους τους ευρωβουλευτές που θα είναι υποψήφοι και σε αυτές τις επόμενες εκλογές. Ευχαριστούμε Εντουάρδο. Και τώρα έχουμε 17 λεπτά περίπου. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από του συναδέλφου να μην υπερβούν τα δύο λεπτά για τα σχολιά τους και τις ερωτήσεις τους. Κλάδια Μοντέρο, παρακαλώ, από το ΕΛΚΑ. Κλάδια, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σε όλους. Επιτρέψτε μου καταρχήν να συγχαρώ όλους όσους ε, συμμετείχαν σε αυτή την τελευταία task force για τον τουρισμό ε, και θέλω να ευχαριστήσω εδώ τον πρόεδρο του τον κύριο Γέλη αλλά και εδώ τους ομιλητές μας μας έκαναν σχετικές παρουσιάσεις 7 λεπτά ο καθένα και λίγο περισσότερο, ω προ τα όσα επέδειχαν στο πλαίσιο αυτή τη τελευταία θεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, και τα όσα λοιπόν επιτέθηκαν εδώ αποτέλεσαν αποτέλεσμα της δέσμευσης που επέδειξαν όλοι όσοι πίστευαν πραγματικά στην αξία του τουρισμού σε αυτή την τελευταία περίοδο. Και αυτό ε, που ε, κάναμε πραγματικά όλοι μας, όπως υπόθηκε, ήταν ε, το να μην συνεχίσουμε με τις δικές μας χωριστέ πολιτικές ατζέντε, έτσι ώστε να δώσουμε την απαραίτητη σημασία σε αυτόν τον κλάδο, ο οποίος πραγματικά είναι τόσο σημαντικός από άποψη ΑΕΠ και από άποψη δημιουργία θέσεων εργασίας και βέβαια ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός και για τις μικρομεσαίες ε, επιχειρήσεις και το πώς μπορούμε να τις υποστηρίξουμε καλύτερα. Όλα λοιπόν ε, τα οποία έγιναν, όλη αυτή η δουλειά που έγινε και για παράδειγμα στο επίπεδο του Μανιφέστο και στο επίπεδο της Task Force θα πρέπει να πω ότι ήταν ε, στις απαρχές τους πολύ δύσκολο να οδηγήσουν σε συγκεκριμένες ενέργειες από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωστόσο, μέσα στα τέσσερα χρόνια που ε, παρήθαν, πράγματι είδαμε τελικά να υπάρχουν συγκεκριμένε προτάσει και συγκεκριμένε δράσει που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επί των οποίων μπορούμε να εργαστούμε. Και ελπίζω ότι στην επόμενη ε, εντολή, στο επόμενο κοινοβούλιο, θα είμαστε ε, σε θέση να συνεχίσουμε αυτή την καλή δουλειά που κάνουμε σε αυτόν τον κλάδο, ειδικότερα όπω αναφέρθηκε προ όφελο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και εδώ αναμένουμε ακριβώ να υπάρξει και περισσότερη υποστήριξη χρηματοδοτική, γιατί όπω είπε και ο κύριο Εντουάντο Σανταντέρ, θα χρειαστούν αυτά τα περιστέρω κονδύλια ακριβώ για να επενδύσουμε στην τεχνολογία, ε, στην ε, ψηφιοποίηση, στου ε, έξυπνου προορισμού, στι έξυπνε ευφυεί πόλει και ούτω καθεξή. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να προωθήσουμε και να αναδείξουμε καλύτερα του τουριστικού προορισμού με βιώσιμο και με ευφυή τρόπο και φυσικά ο, ο κλάδος του τουρισμού συνδέεται άρρηκτα και με τον ε, τομέα των ε, μεταφορών. Και γι' αυτό ακριβώς στο πλαίσιο του τουρισμού, όταν λέμε ότι θέλουμε να προωθήσουμε περισσότερο την κινητικότητα, θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε ακριβώς ε, ο τομέα των μεταφορών να συμβάλλει σε αυτό. Ε, σας ευχαριστώ για μία ακόμα φορά θερμά και νομίζω πραγματικά ότι κάναμε πολύ καλή δουλειά μέχρι στιγμής. Ε, είχαμε μία σειρά από επιτεύγματα και ε, νομίζω πως το επόμενο ε, πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα έχουμε τα καλέτητα απαραίτητα χρηματοδοτικά κονδύλια έτσι ώστε να δώσουμε μία νέα όθηση στην ανάπτυξη του τουρισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Μοντέιρο. Κυρία Ιάλα Σάντερ, έχετε το λόγο. Ναι, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω και να εγκομιάσω το έργο αυτής Task Force ε, αυτήν τη θητεία. Πάντα περιμένει κανείς περισσότερα βέβαια. Ε, πάντα υπάρχουν στιγμές ε, όπου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν αναφέρομαι στην κυρία Ανθρωσοπούλου εδώ που είναι κατά κάποιο τρόπο η ο ανθρωπός μας στην Κομισιόν, αλλά γενικότερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, συχνά δεν έδωσε αρκετή σημασία σε πολιτικό επίπεδο στο θέμα του τουρισμού όταν όλο και πιο πολύ αυτός ο τομέας ε, ουσιαστικά μετατρέπεται σε μια προώθηση της Ευρώπης γενικότερα, μια διαφήμιση της Ευρώπης. Θα έπρεπε λοιπόν να είχαμε επενδύσει περισσότερα στον τουρισμό και στον εσωτερικό τουρισμό, όχι μόνο στον εξωτερικό, έτσι ώστε πολλές από τις προκαταλήψεις που βλέπουμε να αναδύονται αυτή τη στιγμή να μην υπήρχαν. Ε, δύο ερωτήσεις στην κυρία Θανασοπούλου. Ήθελα να ρωτήσω με βάση την ειδική δημοσιονομική γραμμή, την οποία προφανώς και υποστηρίζω, εάν μπορείτε να μας ε, πείτε αν η Κομισιόν, εν πάση έχει κάποιο, κάποιο αριθμητικό στοιχείο να μας δώσει σε ό,τι αφορά τον ευρωπαϊκό προπολογισμό το τι επενδύθηκε απευθεία ε, άμεσα στον τομέα του τουρισμού, τι μπορούμε δηλαδή να ε, πούμε για να συγκρίνουμε. Ε, αν αυτά τα 400 εκατομμύρια είναι αρκετά ή όχι, εμένα μου φαίνονται λίγα. Ε, υπάρχει βέβαια το Invest ε, EU και το προηγούμενο το FC. Εκεί δεν υπήρχε, δεν δόθηκε αρκετή έμφαση στον τουρισμό. Ε, και επίσης θα θέλαμε να ξέρουμε αν υπάρχει κάποιο, ε, αν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με την νομοθεσία, ε, μια χαρτογράφηση αν θέλετε, διότι η νομοθεσία επηρεάζει τον τουρισμό σε μια σειρά από τομείς, ε, αλλά αυτό δεν το έχουμε εμείς ε, ετοιμάσει επαρκώς. Επίσης, οι προτεραιότητες στις οποίες αναφερθήκατε ε, έχουν κάποια σειρά προτεραιότητας μεταξύ τους και πώς συνδέεται αυτό με τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και την στρατηγική 2030 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε κυρία Γιάλα Σέντερ. Κύριε Κράμερ, το λόγο για δύο λεπτά. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για τις παρουσιάσεις σας και για τη δουλειά που κάνατε την τελευταία πενταετία για τον τουρισμό. Ξέρω ότι ήταν δύσκολο το εγχείρημα, αλλά σημαντικό ήταν γιατί τα πράγματα προχώρησαν αργά μένα, αλλά προχωρούν. στα αγγλικά. Η επιτροπή αυτή ονομάζεται Επιτροπή ε, Transport and Tourism, μεταφορών και τουρισμού. Μιλήσαμε λοιπόν για τον τουρισμό. Ε, Λέγοντα «fremdverkehr» στα γερμανικά, είναι ένα όρο που δεν χρησιμοποιούμε πια στα γερμανικά η κυκλοφορία των ξένων. Δηλαδή, έχουμε σταματήσει να λέμε αυτή τη λέξη. Ε, αναφέρομαι στου ε, διερμηνής ε, λέει ο κύριος να λέτε τουρισμός ο τουρισμός λοιπόν είναι ένα σημαντικό πράγμα το είπε και η κυρία Αθανασοπούλου είναι σημαντικό ε, αντιστοιχεί σε 45 δισεκατομμύρια ε, πολλά από τα οποία είναι στον τομέα της κρουαζιέρας για να αναπτύξουμε λοιπόν την κρουαζιέρα, ναι, φτιάχνουμε πολλέ ε, δουλειέ, ε, κοστίζει αντιστοιχεί σε εκατομμύρια. Αλλά για την ποδηλασία, για την τουριστική ποδηλασία, αν βάλουμε 5-10 εκατομμύρια, ε, μα λένε ξαφνικά αυτό δεν είναι εύκολο. Αλλά πάμε και επενδύουμε πάρα πολύ στι κρουαζιέρε. Ξέρετε τι, ε, πρέπει να κάνουμε τα πράγματα πιο ισορροπημένα. Τα πράγματα εξελίσσονται πιο γρήγορα από ό,τι βλέπουμε. Το είδαμε και στη Βιέννη. Εγώ ήμουν ε, σε ένα βιολογικό μοντέλο. Ε, το οποίο, στο οποίο όλες οι δράσεις, ε, όλες οι δραστηριότητες γίνονται με βιώσιμο τρόπο. Μετά έχετε κόσμο που ταξιδεύει με βιώσιμο τρόπο, που δεν πάει κάπου με αυτοκίνητο, για παράδειγμα. Ε, και πάνε και ποδηλάτες που προστατεύουν το περιβάλλον σε τέτοια μοτέλ. Πρέπει λοιπόν να σταματήσουμε να υποστηρίζουμε τα πράγματα που καταστρέφουν τον τουρισμό αλλά να, και τη φύση, αλλά να υποστηρίξουμε τα άλλα. Ε, καμιά φορά μπορεί να είναι πιο ακριβά αυτά, αλλά σίγουρα δεν καταστρέφουν τον τουρισμό. Ο τουρισμό είναι πολύ σημαντικό για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει, ε, αλλά και για τι τοπικέ οικονομίε για τι μεγάλε επιχείρησει δεν είναι κάτι τόσο σημαντικό, αλλά είναι σημαντικό να το προστατεύσουμε. Και εκεί θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για την υποστήριξη που μα έχετε προσφέρει τόσα χρόνια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κράμερ, κυρία Ανάτου. Merci, Madame le Président. Merci. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, σας ευχαριστούμε για τις παρεμβάσεις και για το έργο σας. Οι Βρυξέλλες έχουν αρμοδιότητα υποστηρικτική στον τουρισμό βέβαια, αλλά μου κάνει εντύπωση σε, μια έγγραφος Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων της Κομισιόν για το νέο πλαίσιο του ευρωπαϊκού τουρισμού, μεταξύ των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει αυτός που λέει να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή ηθαγένεια διότι οι ανταλλαγές οι τουριστικές ε, θρέφουν την ευρωπαϊκή ηθαγένεια και την ε, κατανόηση του άλλου. Θέλει η Κομισιό να βασιστεί στον τουρισμό για να προωθήσει το νομοσπονδιακό τη σχέδιο. Ακούστε, η ευρωπαϊκή ηθαγένεια ε, είναι μια έννοια εντελώ αβάσιμη που βασίζεται ουσιαστικά σε ένα νομικό ε, τεχνητό ε, εφεύρημα. Ο κόσμος γνωρίζει την Ευρώπη λόγω των εθνών που την αποτελούν. Και μου έκανε εντύπωση επίσης ότι πέρυσι τελικά η υποψηφιότητα μιας ουγγρικής πόλης δεν ελήφθη υπόψη ε, ως Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Πολιτισμού το 2023 γιατί είπε το, η Επιτροπή Επιλογής ότι το κλιπ ε, το βίντεο κλιπ ε, έκανε προπαγάνδα υπέρ μιας λευκής και χριστιανικής Ευρώπης. Αυτό είναι πραγματικά απίστευτο. Ε, ορισμένα πράγματα λοιπόν, που μας απασχολούν και που πρέπει να κινητοποιήσουν και τις δημόσιες αρχές και τους Ευρωπαίους συθήνοντες. η απασχόληση. Υπάρχουν πολύ σημαντικά προβλήματα ε, στον τομέα της, ε, του τουρισμού, ε, της, ε, της εστίασης όμως ε, ζητούν οι εργοδότες ε, να προσλαμβάνουν πιο πολλούς μετανάστες και βέβαια ενώ μεταξύ η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί ε, προγράμματα ένταξης και η ανεργία ανεβαίνει. Η ασφάλεια των τουριστών πολύ συχνά αυτή διακυβεύεται από σπήρες οι οποίες παραμένουν ατιμόρυτες. Το, η αγοραστική δύναμη των μισέων τάξεων που έχει πληγεί, οι πολιτικές λιτότητας, η ελληνική κυβέρνηση παραδείγματος χάρη έπρεπε να πουλήσει ε, ορισμένες αρχαιότητες μέχρι πρόσφατα. Ε, η συνύπαρξη μεταξύ τουριστών και ηθαγενών στις, ε, και μεταπών τέλο πάντων. Ορισμένε φορέ δημιουργούνται σημαντικά προβλήματα στη Βενετία, στην Πράγα, στη Βαρκελόνη. Ο μαζικό τουρισμό γίνεται ορισμένε φορέ ένα πραγματικό, μια πραγματική πανούκλα και σκέφτομαι ε, τα διάφορα κουρασιερόπλια αλλά και η κακή συμπεριφορά. Ε, των τουριστών συχνά. Συχνά στι πρωτεύουσέ μα επίση βλέπουμε ότι υπάρχουν μπουτίκ οι οποίε είναι άσχημε και όλε οι οποίε πουλούν σουβενίρ ε, χαμηλή ποιότητα που παράγονται στην Ασία. Ε, και ενώ αρχίζουν να ε, αναγκάζονται να κλείσουν ε, πολλές, πολλά μικρά μαγαζιά επειδή είναι πολύ ακριβή, ακριβά τα νίκια στις τουριστικέ περιοχές. Αυτά ήθελα να σα πω. Ευχαριστώ. Η κυρία Ντεμόντε, έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ θα μιλήσω λίγο πιο επικοδομητικά. Είναι ένας σημαντικός οικονομικός κλάδος, τρίτος στη σειρά στην Ευρώπη. Υπενθυμίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισμα ζητώντα κάποια πράγματα, όχι αντιτιθέμενο στον τουρισμό, θα ήταν αστείο. Αυτό που θέλουν οι τουρίστες είναι μεγαλύτερη άνεση. Πρέπει να διατηρήσουμε την Ευρώπη ως πρώτο τουριστικό προορισμό παγκοσμίω. Ε, διευκόλυνση λοιπόν των θεωρήσεων, ε, κατευθείαν πτήσει, υποδοχή. Γι' αυτό λοιπόν η Κομισιόν πρέπει να ε, κάνει περισσότερε προσπάθειε σε θέματα κατάρτιση. Τώρα, όσον αφορά την συνεργατική οικονομία, απευθύνομαι στην Κομισιόν. Υπάρχει κάποια εκτίμηση αντικτύπου για την οικονομία αυτού του τύπου, διότι στις περιοχές με μεγάλη προσέλευση υπάρχει κίνδυνος να μειωθούν ε, τα καταλήμματα που θα είναι διαθέσιμα προς ενοικίαση στους τουρίστες και έτσι μπορεί τελικά να έχει διαφορετικό αποτέλεσμα αυτή η οικονομία η οποία έχει ως στόχο να, καταστήσει, να υποστηρίξει τη γνησιότητα μιας περιοχής. Αυτό με ανησυχεί. Ε, εγώ πιστεύω ότι για την Κομισιόν προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η διατήρηση και η αύξηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Και η δομή θα πρέπει να μεγεθυνθεί. Το έχουμε ζητήσει ήδη. Χρειαζόμαστε περισσότερους ανθρώπους οι οποίοι θα ασχολούνται στον κλάδο του τουρισμού. Πρέπει να διευκολύνουμε και να ε, αυξήσουμε τον ε, τουρισμό ειδική φύσης, ειδικού χαρακτήρα, κάτι που αποκτά όλο και μεγαλύτερη ε, ελκυστικότητα. Οπότε θέλω να ρωτήσω τον Εντουάρδο αυτό. Τι θα μπορούσαμε να προβλέψουμε για το μέλλον, τι είδου δομή θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για τέτοιου ειδικού τύπου ε, τουρισμού. Πέραν αυτό, να πιστεύω ότι ο καθένας πρέπει να κάνει το καθήκον που τον δυστυχεί. Συμφωνώ. Ε, ε αυτή η επιστολή στον Γιούνκερ και εμεί είχαμε στείλει μια επιστολή στον πρόεδρο και δεν λάβαμε απάντηση. Αυτό είναι παράδεκτο, διότι η Κομισιόν κάνει ό,τι κάνει και εμεί ε, οι βουλευτέ κάνουμε ό,τι κάνουμε ο καθένα το καθήκον του, ε, θα πρέπει να κάνει και κάποιο διάλογο ο πρόεδρο με του βουλευτέ. Το ίδιο και τα κράτη-μέλη. Διότι εγώ πιστεύω ότι η αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να μειωθεί, πρέπει να ενταθεί. Διότι αλλιώ μια κατακαιρματισμένη προσέγγιση των κρατών μελών θα είναι κάτι αρκετά αδύναμο στο παγκόσμιο περιβάλλον. Αυτά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ιστφάν, την Πρόεδρο, όλου του συζητητέ, όλου του ομιλητέ ε, για τι παρεμβάσει του. Τέλο, Ελπίζω στην επόμενη θητεία η Task Force να γίνει υποεπιτροπή, διότι χρειάζεται μεγαλύτερη αυτονομία για να καταφέρει να φέρει περισσότερα αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Ντεμόντε. Για να κλείσουμε, ο κύριος Βιμ Βαντεκάμπ. Έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Ε, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ λοιπόν για, την, όλη τη δουλειά που έχει γίνει στον τομέα του τουρισμού και τον ταξιδιωτικό τομέα. Θα ήθελα όμως να θέσω τρία ερωτήματα να κάνω τρία σχόλια. Καταρχήν σε ό,τι αφορά τις θεωρήσεις. Υπάρχουν πραγματικά αυτή τη στιγμή σωστέ διατάξει για τι θεωρήσει. Για παράδειγμα, ένα Ουκρανό ε, τουρίστα προσέρχεται στην Ευρώπη και θέλει να τη διασχίσει ολόκληρη. Έχει αυτή τη δυνατότητα και υπάρχουν μετά πόλεις όπως η Φλωρεντία, η Βενετία, ε, το Άμστερνταμ ε, που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα. Ε, πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα, γιατί είναι σημαντικό να το λάβουμε υπόψη μας, δηλαδή ότι υπάρχει ο τοπικός πληθυσμός ο οποίος υποφέρει από αυτήν την υπερβολική προσέλευση των τουρισμών. Επίσης θα πρέπει να αναλογιστούμε τις, την ποιότητα των θέσεων εργασίας στον κλάδο του τουρισμού, γιατί δεν είναι γνωστός ο κλάδος του τουρισμού για την ποιότητα των θέσεων εργασία του. Δηλαδή, συνήθω αναζητούν ε, νέου, αλλά θα πρέπει να προσφέρονται και οι κατάλληλε θέσει εργασία, καλέ συνθήκε εργασία. Αυτά λοιπόν είναι τα σχόλια που θέλω να κάνω και από την πλευρά μου. Ευχαριστώ. Merci beaucoup, ε, Ευχαριστώ, κύριε Βαντενκάμπ. Και τώρα απευθύνομαι στου ε, ε ομιλητέ. Έχετε λίγο χρόνο όμω για να απαντήσετε, γιατί αργήσαμε. Έχετε καθένα τρία λεπτά, ξέρω ότι είναι λίγα όμως ε, για να έχουμε μια εικόνα ε, να υπάρξουν κάποιες απαντήσεις. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε κυρία Πρόεδρε σε ό,τι αφορά το ερώτημα της κυρίας Αγιάλα για τα αριθμητικά στοιχεία στον προπολογισμό που, που αφορούν τον τον τουρισμό απευθεία. Θα επανέλθουμε και θα σας πούμε πώ ακριβώ διαθέσαμε τον προπολογισμό του κόσμου στον τομέα του τουρισμού. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Σε ό,τι αφορά τώρα το ερώτημα Τη κύρια Ντερμόντε για την συνεργατική οικονομία, κατά πόσο υπάρχει μια μελέτη αντικτύπου. Εδώ θέλω να πω ότι έχουν γίνει μια σειρά από μελέτες ε, σε ό,τι αφορά τους διάφορους τομείς της συνεργατικής οικονομίας και σε ό,τι αφορά τη βραχυπρόθεσμη ε, διαμονή. Έχει γίνει και μια έρευνα ε, γενικότερη για την συνεργατική οικονομία και το μέγεθός της. Κάθε δύο χρόνια υπάρχει το ευρωβαρόμετρο όπου παρακολουθούμε πώς αντιλαμβάνονται οι πολίτες της Ευρώπης στην συνεργατική αυτή οικονομία. Αυτό δεν σημαίνει ότι γνωρίζουμε ότι ε, τα πάντα για αυτό το φαινόμενο το οποίο εξελίσσεται. Θέλουμε να μπορέσουμε λοιπόν να, εντοπίσουμε εστιασμένες μελέτες για τον αντίκτυπο της συνεργατικής οικονομίας ε, ε, στην, στον τομέα της μακροπρόθεσμης διαμονής. Ε, τα ερωτήματα του κ. Κάμπ τώρα για τι θεωρήσει Να θυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάσει την πρότασή τη για το recast, την αναδιατύπωση δηλαδή του, του κώδικα θεωρήσεων. Ε, ε, υπάρχουν βελτιώσεις, χρειάζεται μια ισορροπία μεταξύ ασφάλειας και της ενίσχυση όμως των τουριστικών ροών σε ό,τι αφορά τον υπερβολικό τουρισμό είναι ένα περίπλοκο φαινόμενο αυτό συνδέεται με διάφορες πτυχές εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι απλά θέμα ε, ροών ε, τουριστικών που δεν είναι ισορροπημένες είναι, υπάρχει μια ευρύτερο ζήτημα θα πρέπει ε, να το μελετήσουμε περαιτέρω αποκινούμε τους προορισμούς αυτούς είναι τοπικό το φαινόμενο αυτό θα πρέπει λοιπόν να το συζητήσουμε με τις τοπικές αρχές και τις περιφερειακές αρχές και τις εθνικές αρχές για το θέμα αυτό και, τε, τέλος για τις εθνικές εργασίες είναι αλήθεια ότι η ελκυστικότητα των επαγγελμάτων αυτών στον τουριστικό τομέα είναι ένα ζήτημα υπάρχει βεβαίω και ένα κενό εκεί εργαζόμαστε από αυτού μέσω μελετών μέσω ενό project στα πλαίσια του Blueprint, που διαθέσαμε 5 εκατομμύρια ευρώ στα πλαίσια του Erasmus Plus, για να εξετάσουμε τι ε, ε, προβλέψεις των διαφόρων δεξιοτήτων ε, και βεβαίως ε, κάποια προφίλ εργασίας που συνέχεια οι εθνικές αρχές που είναι υπεύθυνε για το περιεχόμενο της εκπαίδευσης στον τομέα του τουρισμού να μπορούν να αποφελθούν από αυτά. Ε, τέλος να πω ότι τα τελευταία πέντε χρόνια έχουμε δημιουργήσει και ένα ξεχωριστό κλάδο για τον τουρισμό στα πλαίσια του EURES που είναι το Ευρω... η Ευρωπαϊκή Διεκτική Πύλη για την εργασιακή κινητικότητα. Προσπαθούμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε το θέμα των δεξιοτήτων και των συνθήκων εργασίας ε, όσο περισσότερο μπορούμε, λαμβάνοντας υπόψη βέβαια ότι η αρμόδιότητά μας ε, στον τομέα του τουρισμού είναι περιορισμένη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κύριε Σαντάντερ, έχει το λόγο παρακαλώ. Θα μιλήσω ισπανικά τη γλώσσα του Θερβάντες. Η κυρία Γιάλα Σέντερ ε, για τη στόχη τη βιώσιμη ανάπτυξη ε, προφανώ και εγγράφονται στι προτεραιότητέ μα από την αρχή. Από τότε που αναπτύξαμε δηλαδή το μανιφέστο αυτό, ήρθαμε σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Οργάνωση Τουρισμού και βεβαίω ε, πάντα μιλούσαμε για βιωσιμότητα. Είναι προτεραιότητα του μανιφέστο και προφανώς πρέπει να επιμείνουμε κι άλλο και να σεβαστούμε τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Το δεύτερο ερώτημά σας τώρα ε, ποιες θα είναι οι προτεραιότητες για το μέλλον, ε, που θα δώσουμε έμφαση στο τομέα της διακυβέρνησης, διότι όποιος ε, κυβερνάει σωστά κάνει και τα σωστά πράγματα, ε, στον τομέα ε, των δεξιοτήτων. Παρακαλώ, όποιο θέλει να μιλήσει να βγει από την αίθουσα, έτσι, διότι από τη στιγμή απαντάει πυρογνώμονα στα ερωτήματα. Όποιο θέλει να μιλήσει, να βγει. Χρειάζεται λίγο ησυχία ο εμπειρογνώμονό μα για να απαντήσει στα ερωτήματα των συναδέλφων. Συγγνώμη. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Εμέν, επιμένω λοιπόν διακυβέρνηση, δεξιότητες, ε, παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο η εκπαίδευση για το μέλλον του τουρισμού, όχι μόνο του τουρισμού, ε, αλλά και στον τομέα τη πολιτική, Όσο πιο πολλά ξέρουν οι νέοι για τα, για του τουρισμού και όσο περισσότερο ταξιδεύουν, τόσο καλύτεροι άνθρωποι θα γίνουν. Κυρία, κυρία Κράμερ, Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για την ε, θερμή σας υποστήριξη. Η βιωσιμότητα φυσικά και παραμένει μία από τις ε, σημαντικές προτεραιότητες, τις κύριες προτεραιότητες στο πλαίσιο της πρωτοβουλία μας ε, για το μανιφέστο, γιατί χωρίς βιωσιμότητα δεν υπάρχει μέλλον ούτε για μας ούτε για τα παιδιά μας. Ευχαριστώ. Στη γλώσσα του Δάντη, στα Ιταλικά, για να απαντήσω, ο στα Ιταλικά είναι και αυτός που φιλοξενείται και αυτός που φιλοξενεί και αυτή είναι και η βάση του τουρισμού και του μανιφέστου ότι δεν χρειάζεται να αισθάνεται κανεί ότι μονίμω είναι επιχειρηματίε και ότι κάνει μια προσπάθεια για να εξυπηρετήσει κάποιον άλλον να αισθάνεται και ως ε, ε, ε, ε φιλοξενούμενος προέρχεται ο τουρισμός από την λέξη ε, που σημαίνει περιστρέφουμε, τριγυρίζω ε, και για τον κύριο Βαντεκάμπ δεν μιλάω δυστυχώς ε, Ολλανδικά το μόνο που έχω να πω είναι ότι η διεθνοποίηση είναι το μέλλον της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης είναι σημαντικό πράγμα ε, και η Κομισιόν κάνει ό,τι μπορεί. Προσπαθούμε να προωθήσουμε δύο πράγματα για τις ε, θεωρήσεις ε, και για το σχετικό κανονισμό, αλλά έχουμε κάνει σημαντικά βήματα τελευταία και τέλος. Δεν σας ξέχασα. Ευχαριστώ, Κλάουντια. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι το 85% του τουρισμού στην Ευρώπη αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οικογενειακές επιχειρήσεις είναι μικροεπιχειρήσει στην πραγματικότητα και η, Χιου, η Κλάουντια έχει, μας έχει υποστηρίξει πολύ έτσι ώστε δεν έχουν πρόσβαση σε αυτοί που δεν έχουν πρόσβαση σε μεγάλες επιχειρήσεις να μπορούν και αυτοί να βοηθηθούν. Μας βοήθησε πολύ η Κλάουντια, πολλές από τις ενώσεις που προσωπώ εδώ ε, ε, έχουν να κάνουν ακριβώς με μικρές εκμεταλλεύσεις. Ε, ευχαριστώ. Μάλιστα, να ευχαριστούμε τους εμπειρογνώμονές μας που με το λίγο χρόνο που είχαν στη διάθεσή τους απάντησαν στα ερωτήματά σας. Ένας είναι ο στόχος, η Ευρώπη είναι ο πρώτος τουριστικός προορισμός παγκοσμίω, αλλά δεν πρέπει οι ροές αυτές των τουριστών να οδηγήσουν οι πληθυσμοί μας ε, να ζουν πια σε μέρη που έχουν χαλάσει από τον τουρισμό. Πρέπει να μπορούν να αποφεληθούν από αυτόν τον τουρισμό και να γίνει σεβαστή η ζωή των ανθρώπων εκεί. Και βεβαίως ο τουρισμός να είναι ένας μοχλός δράσης για την ανάπτυξη των εδαφών μας, ε, για τον, τη διεθνή έγλη της Ευρώπης, ε, έχουμε και, και πιο πολλούς Κινέζους τουρίστες όπως είπατε, ε, και βεβαίως να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της βιωσιμότητας, διότι η θέρμανση του πλανήτη δεν περιμένει. Σας ευχαριστώ όλους για τις παρεμβάσει Να ευχαριστώ την κυρία Σοπούλου ιδιαίτερα. Και τον κύριο Σανταντέρ. Σας ευχαριστώ πολύ για τις παρεμβάσεις σας. annoncer les résultats dès qu'on a vous dire les copies sont sur table. S'il n'y a pas d'objection, c'est adopté. Allez, nous continuons nos travaux. Συνεχίζουμε τις εργασίες μας. Ε, πριν συνεχίσουμε να θυμίσω το σύνολο των αποφάσεων των συντονιστών ε, σας έχουν ε, μοιραστεί. Ε, εάν δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει κάποια αντίδραση, θα θεωρήσουμε ότι εγκρίνονται. Και ευθύς αμέσως θα δούμε κατά πόσο έχουμε τον κατάλληλο αριθμό για να ψηφίσουμε, αν, έχουμε, αν υπάρχει δηλαδή απαρτία. Αν έχετε η ψηφοφορία, η δοκιμαστική αυτή. Έτσι. Je ferme les Πέρας ψηφοφορίας. Όλα καλά. Ξεκινούμε λοιπόν την πρώτη ψηφοφορία. Σημαντικό το ζήτημα το οποίο εδώ και καιρό το περιμένουμε. Το περιμένουν οι Ευρωπαίοι πολίτες κυρίως. Η πρόταση οδηγίας που βάζει τέλος την αλλαγή του θερινού ωραρίου και που καταργεί την οδηγία 2084. Η κυρία Λούμποκ, λοιπόν, και η έκθεσή της. Θα αρχίσουμε αμέσως. Ξεκινάμε με τρεις παρόμοιε τροπολογίε. Ποιος είναι υπέρ. Όχι, δεν υπάρχει ονομαστική ψηφοφορία. Ζητήθηκε. Μάλιστα il écrit. Λοιπόν, να μην χάνουμε χρόνο. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβασμός 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμό 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμό 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμό 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα Πάμε στο Γιούρι 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ήμκο 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβασμός 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβασμός 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία ΙΤΡΕ 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άγκρι 3. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβασμός 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και πάμε απευθείας στο συμ... στον, στον, στον, 40 ε, με την MV3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Πέττη και Ήμκο λοιπόν εδώ καταπίπτουν και πάμε στο Άγρι 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 43 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές αυτό ευχαριστούμε μας βοηθάει Κράμερ θα το επαληθεύσουμε λοιπόν άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται και περνάμε στο NV4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. NV5 η κυρία Γιάλα Σάντερ λοιπόν επαληθεύσουμε εντάξει NV5 επαληθεύουμε NV4 μάλλον επαληθεύουμε NV4 πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται το NV4 NV5 υπέρ κατά αποχές κύριε Βίμ Βαντεκόρ παρακαλώ συγκεντρωθείτε MV5 εγκρίθηκε MV7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται MV8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και περνάμε απευθείας στο 49 ε, τροπολογία 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 8. Κύριε Βιμ Βαντενκάμπ, θα ψηφίσουμε επί του 49. Άρχεται η ψηφοφορία. Μην ενοχλείτε το τον πλανό σας κύριε Βαντενκάμπ. 49. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Αυτό είχα πει και εγώ. Ήτρε 8. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Ήτρε 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Γιούρι 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα θα ψηφίσουμε επί του συνόλου του κειμένου άρχεται η ψηφοφορία Πέρας ψηφοφορίας. 23 υπέρ, 11 κατά, δεν υπάρχουν αποχές. Η έκθεση λοιπόν αυτή εγκρίνεται και έχουμε πλέον, υπάρχει πλέον θέση του Κοινοβουλίου. Συγχαρητήρια. Allez, nous continuons. Συνεχίζουμε με μια ιδιαίτερη έκθεση για την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που τροποποιεί την ε, οδηγία του Συμβουλίου όσον αφορά τους ειδικού κανόνες ε, για το μέγιστο μήκος των θαλάμων οδήγησης, το οποίο προσφέρει βελτιωμένες αεροδυναμικές επιδόσεις, ενεργειακή απόδοση και επιδόσεις ασφαλείας. Δεν έφτιαξα εγώ τον τίτλο, μην με κοιτάτε έτσι. Η εισηγητής είμαι εγώ, η εισηγήτρια. Οπότε ψηφίζουμε ε, ονομαστική ψηφοφορία γιατί έχουν γίνει διαπραγματεύσεις. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Η έκθεση μου λοιπόν εγκρίνεται με συντριπτική πλειοψηφία. Συνεχίζουμε. Επόμενο σημείο, πρωτόκολλο τροποποίησης της ε, Συμφωνίας ε, εκ για τις θαλασσιέ μεταφορές ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση τη Κροατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση είναι του κυρίου ασή. Καλημέρα κύριε Ασή. Πώς πάτε? Ωραία. Ψηφίζουμε με ονομαστική ψηφοφορία την έκθεσή σας. Άρχεται η ψηφοφορία. Κλείνω την ψηφοφορία τα ίδια. τριπτική πλειοψηφία. Πολύ ωραία. Και τώρα πάμε και συνεχίζουμε με την οδηγία 2008 του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αφορά την διαχείριση των υποδομών, των οδικών υποδομών ε, της κυρίας Αγιούτο. Το θέτουμε σε ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται επίσης με μεγάλη πλειοψηφία. Συνεχίζουμε με το... ενιαία θαλάσσια, την αυθυλιακή Ανία Αθυρίδα. Μεγάλη επιτυχία αυτή η έκθεση. Δική σας κυρία Κλούν. Περνάμε στην τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας. Μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια. Κυρία Κλούν, θέλατε να πείτε κάτι. Θέλετε το λόγο. Θέλετε να πείτε κάτι, κυρία Κλούν. Όχι. Ωραία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τα μέλη τη Επιτροπή, λέει η κυρία Κλούν. Ωραία. Πάμε παρακάτω με το μηχανισμό διασύνδεσης στην Ευρώπη 2014-2020, αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και εγώ είμαι συγγήτρια, άρχεται η ψηφοφορία. Ε, je Πέρας ψηφοφορίας. Δεν χρειάζεται να με φωνάσετε στα ελληνική, κύριε Βαντεκάμπ. Το είδα ότι θα το λέγατε. Λοιπόν... Ε, συνεχίζουμε με την έκθεση του κυρίου Ρικέ για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευση των ναυτικών. Άρχεται η ψηφοφορία. ψηφοφορία. ψηφοφορίας. 32-1 εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Και συνεχίζουμε με τη διασφάλιση βασικής αεροπορικής συνδεσιμότητας ε, ε, όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Τελίτσκα είναι ο εισηγητής, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 31 υπέρ εγκρίνεται. Και τέλος, η διασφάλιση βασικής συνδεσιμότητας των οδικών με εμπορευματικών μεταφορών όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση. Έκθεση της κυρίας Ιζαμπέλα Ντεμόντε, της ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια Κύριε Αντεμόντε. Και τελειώσαμε με τις ψηφοφορίες. Σας ευχαριστώ όλους. Τελειώσαμε. Και τώρα θα περάσουμε στο επόμενο σημείο. Α, όχι. Έχουμε κάποιο χρόνο και θα κάνουμε ένα δεκάλεπτο διάλειμμα. Και όταν επανέλθουμε θα δούμε το σχέδιο καταξιδότηση πράξη σχετικά με τις προδιαγραφές για τα συνεργατικά και ευφύ συστήματα μεταφορών με τον εισηγητή μας, την εισηγήτριά μας και την κυρία Μάισνερ. Κάνουμε διάλειμμα για 10 λεπτά.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

chers collègues, nous allons reprendre nos... Αγαπητοί συνάδελφοι, ξαναρχίζουμε τι εργασίε μα. Ε, για δεν έχετε αντίρρηση. Ξεκινούμε, επαναλαμβάνω, εκ νέου τι εργασίε μα και περνάμε στο σημείο 14 τη μέσα διάταξη. σχέδιο πράξη κατεξιοδότηση για τι προδιαγραφέ. Παρακαλώ, όποιος θέλει να μιλήσει εκτός αίθουσας. Λοιπόν, σημείο 14. Θα εξετάσουμε το σχέδιο πράξη δεξιοδότηση για τις ε, προδιαγραφές των συστήματων έξυπνων μεταφορών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύντομα θα εγκρίνει μια πράξη κατεξιοδότηση για αυτά τα συστήματα έξυπνων συνεργατικών μεταφορών το Κοινοβούλιο έχει ήδη εκφραστεί από αυτού με την της πρωτοβουλία του κύριου Ουέλγη για τη στρατηγική, ευρωπαϊκή στρατηγική σχετικά με το CITS και μετά την τελευταία μας συζήτηση στις 29 Ιανουαρίου πολλά ζητήματα, πολλά ερωτήματα τέθηκαν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τα μέλη μας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε γραπτός που σας εστάλει σε όλους εσάς την περασμένη Παρασκευή. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η διαδικασία παρακολούθησης, εποπτείας, σκρούτινη. Το Κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται για το περιεχόμενο των πράξεων του για να μπορέσει να ασκήσει πλήρως τον ελεκτικό του ρόλο. Και βεβαίως έχει μια περίοδο δύο μηνών για να υποβάλει ενδεχόμενη, ενδεχόμενη αντίρρηση. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει σαφείς πληροφορίες για το ζήτημα και κυρίως να διευκρινίσει πότε η κατεξοδότηση πράξη θα εγκριθεί επισήμως και θα διαβαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα δώσω το λόγο λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρώτα, στην κυρία Κλέρ Ντεπρέ που είναι μαζί μας σήμερα και στη συνέχεια θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια, την κυρία Μάισνερ. Και βεβαίως μετά ξεκινάει η συζήτηση. Κυρία Ντεπρέ, έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που δίνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην, στα μέλη τη Επιτροπής Μεταφορών το χρόνο να εξετάσουν αυτό το σημαντικό ζήτημα. Μιλάμε για έξυπνα συνεργατικά συστήματα μεταφορών ε, και μιλάμε όντω για ένα μελλοντική, μια μελλοντική πράξη εξουδότηση. Από τις, ε, την προηγούμενη ανταλλαγή απόψεων για το θέμα αυτό το Μάιο, τον Ιανουάριο συγγνώμη φέτο, ε, υπάρχει, φαίνεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον για το θέμα αυτό. Και επειδή έχω ασχοληθεί και εγώ μου λεπτομερώς με το ζήτημα, χαίρομαι γι' αυτό. Ε, υπάρχουν, υπάρχει ανάγκη μεγαλύτερων ε, διευκρινήσεων, γι' αυτό και ζητάτε κάποιες περαιτέρω πληροφορίες. Ε, ε μας το ζητήσατε μάλλον γραπτός, απαντήσαμε την προηγουμένη Παρασκευή, με καθυστέρηση βέβαια και λυπάμαι γι' αυτό. Ελπίζω ότι η λαγή απόψεων μας σήμερα να μας βοηθήσει να διευκρινίσουμε περαιτέρω ε, τα ζητήματα αυτά, να εμβαθύνουμε τις γνώσεις μας και την κατανόησή μας και αν υπάρχει οποιοδήποτε περαιτέρω ερώτημα είμαστε εδώ για να απαντήσουμε. Ε, θα ήθελα να ξεκινήσω με την πρώτη διαφάνεια που έχουμε ε, ετοιμάσει. Να σας εξηγήσω λίγο ποιο είναι το πλαίσιο, το ιστορικό, γιατί οι υπηρεσίε της Κομισιόν έχουν ενεργοποιηθεί για το ζήτημα αυτό. Ε, δεν θα εκπλαγείτε δεν θα εκπλαγείτε αν σας πω ότι συνδέεται έντονα το ζήτημα αυτό με το ζήτημα της οδικής ασφάλειας. Εδώ βλέπετε ένα γράφημα το οποίο το γνωρίζετε. Είναι η εξέλιξη σε ό,τι αφορά τα θύματα οδικών ατυχημάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, η ατζέντα μας σε ό,τι αφορά την προσπάθεια μείωσης των θυμάτων και την ασφάλεια των οδικού δικτύου ε, βλέπουμε ότι αυτή η προσπάθεια σιγά σιγά ε, δεν αποδίδει. Δηλαδή δεν έχουμε πια τόσο μεγάλη βελτίωση σε ό,τι αφορά την ασφάλεια στους δρόμους. Δεν μιλάω καν για, τα, για τους σοβαρά τραυματίες ε, όπου είναι πενταπλάσια τα αριθμητικά στοιχεία. Επίσης ε, δεν είναι τυχαίο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ε, ενεργοποιηθεί στο ζήτημα τη οδικής ασφάλειας, έχουν υποβληθεί μέτρα και στα πλαίσια του τρίτου πακέτου κινητικότητα, προσπαθώντα να προσφέρουμε μια απάντηση σήμερα. Το σχέδιο δράσης για την οδική ασφάλεια, κάποια μέλη άλλωστε ασχολούνται ιδιαίτερα με αυτό, φτάνει σε ορισμένα πολύ συγκεκριμένα μέτρα, με στόχο να είναι πιο ασφαλή οι δρόμοι, να είναι πιο ασφαλή τα οχήματα, αλλά και η διάδραση μεταξύ του οχήμα, των οχημάτων αλλά και μεταξύ των, των, του και του δρόμου να είναι ασφαλέστερη. Όλα αυτά αποτελούν μέρος της λύσης. Το CITS, το οποίο όπως το, ονομάζουμε, υπάρχουν πολλοί και διάφοροι τρόποι να αντιμετωπίσουμε την οδική ασφάλεια. Μπορούμε να έχουμε παθητική, ενεργητική οδική ασφάλεια. Εμεί θέλουμε μια συνεργατική οδική ασφάλεια. Κάτι που δεν έχει γίνει ακόμα. Που γίνεται για πρώτη φορά. Ο στόχος της κατεξοδότησης πράξης ε, αυτό που θα ήθελα να πω πρώτα απ' όλα μάλλον είναι ότι το CITS και αυτή η ανακοίνωση, η επικοινωνία μάλλον μεταξύ του οχήματο και της υποδομής που το, και του χρήστη ουσιαστικά εμπίπτει ε, στην οδηγία CITS συνάδελφος που ασχολείται με αυτό δεν είναι εδώ σήμερα. Είναι πάντως ε, ένα από τα αποτελέσματα των εργασιών μας στα πλαίσια της οδηγίας CITS. Τι θέλουμε λοιπόν να πετύχουμε με αυτά τα μέτρα υπό προπαρασκευή. Πρώτα απ' όλα θέλουμε να υπάρχει μια νομική ασφάλεια. Ε, θέλουμε να έχουμε μέγιστη νομική, ε, οδική ασφάλεια θα φτάσουμε, θα φτάσει το μέγιστο επίπεδο αποτελεσματικό του CITS εφόσον όλοι οι, οι χρήστες του οδικού δικτύου θα μπορούν να, να έχουν μια διάδραση μεταξύ τους. Μέσω τη πράξη εξουδότηση, λοιπόν, ε, θέτουμε τι προποθέσει για να συμβεί κάτι τέτοιο. Θέλουμε επίση να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει εμπιστοσύνη στην επικοινωνία αυτή. Βεβαίω και θέλουμε να είναι όλοι συνδεδεμένοι μεταξύ του, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι ο χρήστης, οι χρήστε μπορούν να πιστεύονται μεν του. Δεν χρειάζονται λοιπόν μια σειρά από απαιτήσει ε, στον κανονισμό, ε, προδιαγραφέ που έχουν να κάνουν ακριβώ με το θέμα τη ασφάλεια. Επίση θέλουμε να επιταχύνουμε την εναρμονισμένη προσφορά, εναρμονισμένη μάλλον ευρωπαϊκή ανάπτυξη των υπηρεσιών αυτών για να μην υπάρχει κατακρεματισμός. Επίσης θέλουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για μαζική ανάπτυξη του CIT στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κάτι που δεν έχει συμβεί αλλού και είναι κάτι που θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και του κλάδου μας, του βιομηχανικού. Του βιομηχανικού. Πώς θα το κάνουμε λοιπόν αυτό. Εδώ η βάση είναι η εξής. Θέλουμε όριμες υπηρεσίες να προσφέρουμε, να γνωρίζουμε τι προσδοκάται από εμάς. Αυτή η βάση θα επεκταθεί, θα εξελιχθεί. Γι' αυτό υπάρχουν, θα υπάρξουν πολλαπλές ε, τροποποιήσεις του κανονισμού και βελτιώσεις για να προσθέσουμε υπηρεσίε Να έχουμε όσο γίνεται περισσότερε υπηρεσίε. Ξεκινάμε με ένα περιορισμένο αριθμό υπηρεσιών που όμως θα αυξηθεί. Ήδη προχωρούν οι εργασίες στον κλάδο, σε επίπεδο κρατών μελών, για να υπάρξει περαιτέρω εναρμόνιση περαιτέρω υπηρεσιών που θα καλυφθούν από αυτήν την καταξιδότηση πράξη. Και θα εξετάσουμε τις υπηρεσίες CITS και για την ε, οδήγηση, την ε, μεταφορά χωρίς οδηγό. Ε, θέλουμε να εκμελευτούμε βεβαίω τι νέε τεχνολογίε, αλλά και το υπάρχει, την υπάρχουσα κάλυψη του δικτύου. Είμαστε ανοιχτοί στι νέε τεχνολογίε. Το σημείο αφιτηρία σήμερα ε, θα εξελιχθεί στο μέλλον. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ε, βεβαίω πάντα συμβατότητα με την βάση, με τα βασικά. Πρέπει να μπορούν όλοι να να επικοινωνούν με όλους. Υπάρχει το σημείο της νομικής ασφάλειας που είναι κρίσιμο, ε, αυξημένη ανάπτυξη, να είναι όλοι συνδεδεμένοι με όλους και να υπάρξει συνέχεια στην παροχή της υπηρεσίας. Και πάμε τώρα στην επόμενη διαφάνεια. Ρωτήσατε στην τελευταία ανταλλαγή απόψεων, στήσατε κάποιες πληροφορίες για την ίδια την τεχνολογία. Εμείς επικεντρωνόμαστε σε μεγάλο βαθμό στη διαλειτουργικότητα και η διαλειτουργικότητα ήταν ο στόχο ένα από του στόχου ε, και τη οδηγία και τη πράσινης ταξιοδότηση. Επίση εξηγήσαμε ότι οι τεχνολογίε είναι συμπληρωματικέ. Αυτά τις γραμμέ που βλέπετε εδώ μπροστά σα αποτελούν μέρος ε, της ε, γραψής συνεισφορά που σα στείλαμε, αυτέ αυτές διαφάνειε. Ελπίζω με αυτό το γράφημα να, να καταλάβετε, να διευκρινίσουμε κάπως τα πράγματα. Η πράσινη αξιοδότηση δεν παρεμποδίζει την υπάρχουσα παροχή υπηρεσιών. Ούτε το, το 3G, ούτε το 4G, ούτε το 5G και τα λοιπά δίκτυα. Η πράξη κατοξιδότηση θέλει να ε, επεκτείνει ε, την τεχνολογική αυτή προσέγγιση. Να πω και δύο λόγια τώρα για την προστασία των δεδομένων, γιατί και αυτό συζητήθηκε την περασμένη φορά. Πρέπει να σας πω ότι αυτό το μέτρο δεν μπορεί να παράσχει νομική ασφάλεια σε ό,τι αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Δεν είναι ε, ένα κείμενο που έχει σχέση με την προστασία δεδομένων. Το γενικό πλαίσιο προστασία δεδομένων είναι γνωστό και οι διατάξεις τους ε, εφαρμόζονται κατά γράμμα. Η πράσινη τοξιοδότηση, σε ό,τι αφορά τις απαιτήσει ε, για την ασφάλεια, ε, συνεισφέρει ώστε να, έχουμε, να χρησιμοποιούνται ψευδόνυμα Ελαχιστοποιείται λοιπόν η περίπτωση κακής χρήσης των δεδομένων αυτών. Έχουμε συνεργαστεί στενά με τους συναδέλφους της δικαιοσύνη της αρχής προστασίας δεδομένων, ε, με την, ε, το, το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων ε, και θα λάβουν χώρα διαβουλεύσεις επ' αυτού και στο μέλλον, επισήμως. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ σε κάποια στοιχεία στα οποία ε, προέκυψαν στην περασμένη συζήτηση και να δώσω κάποιες διευκρινήσεις που ίσως να χρειάζονται Το πρώτο που θα ήθελα να πω κάποιοι από εσά αντέδρασαν στο ό,τι αφορά τη σύνθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων. Επ' αυτού πραγματικά να σας πω ότι ποτέ δεν ήταν πρόθεσή μας να είμαστε αχρίαστα περιοριστικοί. Το αντιμετωπίσαμε το θέμα αυτό στις εργασίες μας, ε, διευκρινίσαμε το κείμενο έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία παρανόηση. Δεύτερον, θα πρέπει η πράξη οξυδότηση να είναι ανθεκτική ε, στο μέλλον και να υπάρχει μεγαλύτερη αναθεώρηση. Είχατε μια ανησυχία, ε, εν πάση ρωτήσατε για τη σχέση μεταξύ της πράσινης εξοδότησης και της εξελίξης με το 5G. Εδώ θέλω να υπογραμμίσω ότι πάντα είχαμε εμεί μεγαλύτερη αναθεώρηση στο κείμενό μας για να αντιμετωπίσουμε την συμπερίληψη νέων τεχνολογιών. Και τώρα δίνουμε περισσότερα στοιχεία για τη διαδικασία αυτή. Για την ασφάλεια. Έχουμε διευκρινίσει τη διάδραση μεταξύ αυτού του μέτρου, την προσωρινή ασφάλεια αυτού του μέτρου και τις άλλες ε, νομοθεσίες περί κυβερνοασφάλειας έτσι είναι σαφέστερο πλέον ότι είναι διαφορετικά τα νομικά πλαίσια τα οποία όλα μαζί είναι συμπληρωματικά και έχουν σκοπό να, οδηγηθούν, να οδηγήσουν στο ίδιο αποτέλεσμα. Τελειώνοντας, να πω δύο λόγια ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεγάλη βούληση για να υπάρξει μια μαζική ανάπτυξη του CITS και στα κρατημέλη και στον κλάδο και αυτό με επαναφέρει στην αρχική μου διαφάνεια για την ε, οδική ασφάλεια. Υπάρχει λόγος που είναι κρίσιμη η ανάγκη για αυτή την πράξη του ΣΥΔΟΣ αυτή τη στιγμή. Ελπίζω αυτή η διευκρίνηση, η γραπτή αλλά και η σημερινή μας συζήτηση να σας βοηθήσει να καταλάβετε καλύτερα το τι διακυβεύεται εδώ με την, πράξη, με την κατεξοδότηση πράξη. Είμαστε εδώ για να σας δώσουμε οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία θέλετε και για να απαντήσω στο αίτημα τη κυρία Ντέλη για το χρονοδιάγραμμα η πράξη εξοδότηση θα την έχετε στις 13 Μαρτίου όταν θα είναι διαθέσιμε και όλες οι μεταφράσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να μην μακρηγόρησα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ντεπρέ για αυτές τις εξηγήσει. Δίνω το λόγο στην εισηγήτρια την κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε την Επιτροπή για αυτή την παρουσίαση και όχι μόνο για τη σημερινή παρουσίαση αλλά για τις εκτενείς πληροφορίες που μας έχει διαθέσει. Μα αποστήλατε δηλαδή κάποια έγγραφα. Ε, βέβαια θα ήθελα να τα είχαμε λάβει λίγο νωρίτερα από το που μα τα στείλατε, αλλά σε κάθε περίπτωση είχα δυνατότητα να τα κοιτάξω, αν και όχι εντελώ. Σε κάθε περίπτωση, εγώ έχω ήδη αναφέρει ότι ναι, υποστηρίζω αυτή την κατεξουζότηση πράξη και το λέω ευθύ εξ αρχή. Γιατί υπήρξαν ε, και πολλά ε, αντίθετα επιχείρηματα που εκφράστηκαν κατά τελευταία συζήτηση που έγινε και τα έλαβα πολύ σοβαρά υπόψη μου και στο πλαίσιο αυτή τη συζήτηση έχω ε, εξετάσει και προσεκτικά τα διάφορα έγγραφα. Σε κάθε περίπτωση, θεωρώ πω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει αυτό την οποία καλέσαμε να κάνει. Ε, δηλαδή είχαμε και την έκθεση από την πλευρά του συναδέλφου Γιουλέβη, όπου ε, αναφερόταν ότι θέλουμε να προωθήσουμε την καινοτομία και στις οδικές μεταφορές. Ναι. Ε, και αν, αν θυμάμαι καλά, αυτέ τι ιδέε που είχαν εκφραστεί από την πλευρά των φιλελευθέρων τι έχουμε υιοθετήσει και εμεί. Άρα λοιπόν, αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε πώ μπορούμε να δώσουμε μια συνέχεια σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί η Επιτροπή νομίζω πω έχει δίκιο σε αυτό που προτείνει, ότι δηλαδή ε, θέλουμε να υπάρξει κατεξουσιοδότηση πράξη όταν θα έχει εδραιωθεί επαρκώ η σχετική τεχνολογία. Για παράδειγμα, το 5G έχει προχωρήσει αρκετά, αλλά δεν είναι ακόμα αρκετό όριμο, δεν έχει αντρεωθεί ακόμα. Δηλαδή, πολλοί λένε ότι στα τέλη του ε, έτου ε, θα χρησιμοποιείται. Αλλά αν περιμένουμε μέχρι τα τέλη του έτου, τότε αναμένουμε ουσιαστικά το νέο ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και υπάρχει ο κίνδυνο ενώ σε αυτή την περίπτωση να μην βελτιωθεί μια κατάσταση την οποία θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε από τώρα. Γι' αυτό και ανέφερα κατά τελευταία συζήτηση ότι η δική μα τοποθέτηση και η σχετική απόφαση θα πρέπει να είναι ουδέτερη σε ό,τι αφορά την τεχνολογία. Εάν όμω υπάρχουν μόνο δύο τεχνολογίε σε ένα κλάδο, εκ των οποίων η μία ακόμα δεν είναι διαθέσιμη, τότε τα πράγματα είναι ξεκάθαρα και δεν υπάρχει μεγάλο δίλημα δηλαδή στην απόφασή μα. Αναφέρθηκε και η ανάγκη τη συμβατότητα. Εδώ εγώ ασχολήθηκα με τι τεχνικέ λεπτομέρειε, οπότε δεν θέλουμε να δώσουμε ε, το, το λανθασμένο την λαθασμένη εντύπωση. Δηλαδή το θέμα με το 5G από ό,τι κατάλαβα ε, βρίσκεται στο latency, δηλαδή τη μικρή καθυστέρηση σε ό,τι αφορά τη διαβίβαση των δεδομένων. Ε, αλλά νομίζω πως αυτό διορθώνεται και νομίζω πως ε, ε, με την τεχνολογική εξέλιξη που βιώνουμε αυτή την περίοδο και αφού η Επιτροπή μας λέει ότι σε κάθε περίπτωση το σύστημα θα ενσωματώσει στο μέλλον και το 5G δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε ό,τι αφορά δηλαδή την επικοινωνία αν θέλετε συμβατότητα μεταξύ των δύο διαφορετικών συστημάτων στο μέλλον. Ε, και αυτή η ρήτρα αναθεώρηση που περιλαμβάνουμε ακριβώ αυτό ε, διασφαλίζει. Ότι δηλαδή μόλι υπάρξει νέα τεχνολογία θα πρέπει να ενσωματώνεται και αυτή στο σύστημα. Και νομίζω πω αυτή είναι και μόνη άγουσα που μπορούμε να ακολουθήσουμε. Δηλαδή οι τεχνολογικέ ε, εξελίξει θα πρέπει, ε, επειδή ακριβώς είναι τόσο ραχδές να τις λαμβάνουμε ε, υπόψη μας ε, ό,τι μπορούμε, αλλά δεν μπορούμε δηλαδή να προδικάσουμε τι θα έχουν αναπτύξει μέσα σε τρία χρόνια οι ερευνητέ. Άρα λοιπόν αυτό που κάνουμε είναι να υιοθετούμε την τεχνολογία που υπάρχει αυτή τη στιγμή διαθέσιμη και από εκεί και μετά να έχει επαρκώ ανοιχτό χαρακτήρα το σύστημα για να ενσωματώσει μελλοντικέ τεχνολογίε. Και νομίζω πω αυτό είναι και το ε, και, το, και αυτό που προτείνουμε και αυτό είναι το μόνο δυνατό και νομίζω πως ε, ακόμα και αν ακολουθήσουμε τη, τη σωστή, το σωστό χρονοδιάγραμμα θα έχουμε μόνο ένα μήνα πριν από την εκλογή του νέου κοινοβουλίου για να περάσει αυτή η πρόταση οπότε ελπίζω να τα καταφέρουμε γνωρίζω βέβαια πως υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι δεν ε, συμφωνούν με τις δικές μου απόψεις υπάρχουν και βέβαια και κάποια οικονομικά συμφέροντα υπάρχουν και κάποιες περιφερειακού χαρακτήρα προτεραιότητες ε, πάντως εγώ ως Ευρωπαία νομίζω πως αυτή είναι σωστή λύση δηλαδή ως Γερμανίδα ενδεχομένω να είχα διαφορετική άποψη αλλά νομίζω αν το δούμε από την ευρωπαϊκή οπτική γωνία θα πρέπει να το προωθήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριο Βίμ Βαντεπάνκ. Έχετε το, ε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ήθελα να πω ότι σε μεγάλο βαθμό συμφωνώ με την κυρία Μάισνερ, την εισηγήτρια. Ε, σε μικροπράγματα όμως έχουμε κάποιες διαφορές. Σε μικρολεπτομέρειες ε, και πιστεύω ότι αυτές τις λεπτομέρειες πρέπει να τις δούμε με προσοχή. Συμφωνώ με τη Ζεζίν και ευχαριστώ την ε, Επιτροπή για όλες τις πληροφορίες. Μας ε, παρουσίασε πολύ λογικά τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να προσέξουμε και τι δεν πρέπει να προσέξουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή μπροστά μας έχουμε ένα non-paper, αυτό έχουμε λάβει. Τι νομική ισχύ έχει ένα non-paper. Αν πάω στην παράγραφο στη σελίδα 7 όπου λέει ότι ε, αυτή η κατεξιοδότηση πράξη αναφέρει ότι θα περιμένουμε το 5G και ότι αυτό θα ενισχύσει ε, την υπερασπίση της υπόθεση Η Κομισιόν λέει όχι, ε, ότι αυτό συγγνώμη, θα είναι αρνητικό. Η Κομισιόν λέει το αντίθετο, ότι θα είναι θετική η εξέλιξη για το 5G. Και η, η ερώτησή μου προς την Κομισιόν είναι τελικά ποια είναι η νομική ισχύ αυτού του non-paper. Μπορούμε να αναφερόμαστε στο μέλλον σε αυτό το έγγραφο ή όχι. Και από άψη βιομηχανική ε, ανάπτυξη ήθελα να το καταλάβω. Και μετά κάτι άλλο. Ε, δεν είμαι βέβαιο αν κατάλαβα καλά αφορά και τα όσα είπε ο κ. Κόχ. Όλο αυτό το CITS μου φαίνεται πολύ πιο ευρύ από απλά τα θέματα οδικής ασφάλειας. Αφορά το μέλλον, την ε, ανάπτυξη αυτόνομων οχημάτων με όλες ε, τις ε, συνδέσεις που θα χρειαστούν στο μέλλον. Όταν μας λέει λοιπόν η Κομισιόν ότι το CITS αφορά την οδική ασφάλεια, και γι' αυτό πρέπει να έχουμε αυτή την τεχνολογία την ασύρματη. Ναι, συμφωνώ. Αλλά έχουμε πολύ ευρύτερε και μεγαλύτερε εξελίξει αυτή την εποχή. Και εδώ έρχομαι στο πιο σημαντικό μου ερώτημα. Δηλαδή, πόσο σημαντικό είναι το άρθρο 33 και κυρίως ποια είναι η σχετική διαδικασία. Ε, το είπε και η κυρία Μάισνερ και η κυρία Ντεπρέ. Οι νέες τεχνολογίες θα έρθουν κάποια στιγμή. Ωστόσο, ο τρόπος, ε, ή μάλλον ε, ε, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα βάσει του οποίου θα αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν το γνωρίζουμε, δεν το μαθαίνουμε από πουθενά. Και γι' αυτό διαφωνώ με την κυρία Μάισνερ. τι θα κάνουμε τώρα, πώς θα δράσουμε γρήγορα και με τον κατάλληλο τρόπο. Η κυρία Μάισνερ λέει εντός έξι μηνών Και όμω αυτέ οι τεχνολογίε υπάρχουν ήδη. Όλα τα θέματα συμβατότητα, λειτουργικότητα υπάρχουν ήδη ω προβλήματα. Και κάτι τελευταίο, κυρία Πρόεδρε. Μα φαίνεται αστείο που λέει ότι αυτή η προσέγγιση ε, δεν είναι περίπλοκη τεχνολογικά και έτσι επιλέγουμε το wireless. Δεν είναι ουδέτερη τεχνολογικά. με ποια διαδικασία θα εντάξουμε το 5 σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή την κατεξοδότηση πράξη. Και μετά λάβαμε μία επιστολή από το EUTP, τον φορέα μεταφορών στην Ευρώπη, και αυτοί μα ζητούν, και το λέω στα αγγλικά, μα ζητούν να δώσουμε προσοχή στην ανακοίνωση στο Communication Control Based Command, το λέω στα αγγλικά. Αστικές, υπεραστικές εφαρμογές για τις ιδεοδρομικές μεταφορές. Ζητώ λοιπόν από την Κομισιόν τι θα κάνουμε με αυτή την τεχνολογία και στο πλαίσιο του 5G και πώς θα εντάξουμε μια ε, ε, ε, μονομερή επιλογή του wireless και τι θα γίνει με τη διαδικασία του άρθρου 33. Αυτά. Ευχαριστώ κύριο Σχέρτουγκ. Ε, σας ευχαριστώ πολύ και εξ ονόματος της ε, Σοσιαλιστικής Ομάδας ε, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, καταρχήν, από τις αρχές θα ήθελα να πω ότι πάντοτε προτεραιότητα θα πρέπει να δίνουμε στην λεπτομερή εξέταση ε, των ζητημάτων Ε, από ότι η ταχύτητα σε ό,τι αφορά την άγουσα. Άρα νομίζω και με βάση νομίζω και ένα ε, ε, πρόσφατο νέο δυστύχημα που είχαμε στις Ηνωμένε Πολιτείε, θεωρώ πως από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακολουθούμε τη σωστή διαδικασία. Δηλαδή εξετάζουμε τα πάντα διεξοδικά για να μην έχουμε απώλεια ανθρωπινών ζώων. Από εκεί και μετά συμφωνώ με τα όσα είπε η συνάδελφος Μάισνε. το άρτυπο, ανεπίσημο αυτό έγγραφο δεν το έχω ακόμα νόσω, οπότε δεν μπορώ ακόμα να το εκτιμήσω, αλλά τα όσα έχω δει μέχρι στιγμής νομίζω καταδεικνύουν ότι μπορούμε να κάνουμε μια πραγματική διαφοροποίηση ανάμεσα στο μικρής εμβέλειας και μεγάλης εμβέλειας, short range και long range. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι η τεχνολογία η οποία υπάρχει διαθέσιμη σήμερα και χρησιμοποιείται μπορεί να ε, δοκιμα... να, να χρησιμοποιηθεί πλέον και εκτό δοκιμών. Ε, και νομίζω πως και ο, ο κλάδος αναμένει αυτό και όχι μόνο ο κλάδος, αλλά ε, και παγκοσμίω δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι βρισκόμαστε σε ανταγωνισμό με άλλε περιοχέ του κόσμου, με άλλε χώρε. Οπότε νομίζω πω θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τα όσα ήδη έχουμε στη διάθεσή μα και να μην καθυστερούμε την όλη διαδικασία τεχνητά. Από την άλλη βέβαια πλευρά θα πρέπει να είναι δυνατό να διασφαλιστεί εν λόγω συμβατότητα, δηλαδή αυτή ακριβώς η ουδετερότητα σε ό,τι αφορά τις χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες όταν θα είναι πλέον ε, ευρύτατα διαθέσιμη η νέα, για παράδειγμα, τεχνολογία 5G. Ε, και από εκεί και μετά θα πρέπει να διασφαλίσετε και το backwards compatibility, δηλαδή η συμβατότητα προς τα πίσω. Δηλαδή ε, τα οχήματα, Δηλαδή, τα οποία δεν έχουν ακόμα μια τέτοια τεχνολογία να είναι δυνατόν να εξοπλιστούν με αυτήν εκ των υστέρων. Γιατί είναι σημαντικό στο πλαίσιο της εφαρμογής αυτών των τεχνολογιών στην, ε, στο δρόμο, στις οδικές μεταφορές, να χρησιμοποιούνται από όλους. Δηλαδή δεν θα ήθελα να φτάσουμε σε μια κατάσταση όπου η εικόνα θα είναι μεικτή. Δηλαδή θα έχουμε ένα ε, τμήμα των οχημάτων τα οποία δεν θα είναι συμβατά και κάποια που θα είναι. Δηλαδή να μην υπάρχει τελικά μια τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί και η οποία θα είναι μόνο διαθέσιμη για τα νέα οχήματα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την προσέγγιση ότι να αξιοποιήσουμε δηλαδή την ήδη διαθέσιμη τεχνολογία ε, και νομίζω ε, πως και βραχυπρόθεσμα πρόθεσμα θα πρέπει να είναι δυνατόν στους Αυτοκινητόδρομου να καταστήσουμε διαθέσιμη τη δυνατότητα αυτόματη οδηγήση. Νομίζω ε, πως εδώ αξίζει να αναφερθούμε ότι υπάρχει μια δοκιμαστική φάση στους γερμανικού αυτοκινητόδρομού εδώ και δύο χρόνια, η οποία κατά τη δική μου άποψη ε, ήδη έχει καλά αποτελέσματα και, το, ε, και από την οποία μπορούμε να αντίσουμε και κάποια διδάγματα. Ε, από εκεί και μετά αναμένουμε ενδιαφέρον την επόμενη συζήτηση που θα κάνουμε όταν θα έχουμε διαβάσει ε, εντελεχώ αυτό το έγγραφο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Στο πλαίσιο πάντω τη εν λόγω πρωτοβουλία θα πρέπει να διασφαλίσουμε την ουδετερότητα σε σχέση με τι τεχνολογίε. Χωρί όμω αυτό να σημαίνει ότι θα πρέπει να ε, καθυστερήσουμε την όλη διαδικασία. Κατά τα λοιπά ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατάρτιση αυτού του εγγράφου και τι προσπάθειε που έχει κάνει μέχρι τώρα. Ευχαριστώ, κύριο κύριος Ρικέ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίαση και για τα έγγραφα που μας μοίρασε. Όταν είχαμε για πρώτη φορά μάθει για αυτήν την πράξη δεξιοδότηση, είχα εκπλαγεί και ρώτησα εάν αυτή η πρόταση κρύβει κάποια πράγματα. Ε, ε, έκτοτε μελέτησα, συνάντησα και την Κομισιόν, παραμένω εξαιρετικά επιφυλακτικός. Έχω αντιρρήσεις και επί των τύπου, επί της διαδικασίας, αλλά και επί της ουσίας. Βεβαίως, εντάξει, ο στόχος της ασφάλειας που θέτει η Κομισιόν, κανείς δεν έχει αντίρρηση προφανώς. Όλοι θέλουμε να βελτιώσουμε την ασφάλεια και να χρησιμοποιήσουμε τις τεχνολογίες που το επιτρέπουν αυτό. Εδώ συμφωνούμε. Μπαίνουν κάποια ζητήματα όμως πρώτα επί των τύπων, έτσι. Ένα γενικότερο ζήτημα. Οι οδηγίες CITS που τροποποιείται εδώ με μια εκτελεστική πράξη είπατε ότι θα πρέπει να προβλέψουμε και άλλες πολλές εκτελεστικές πράξεις στο μέλλον. Ε, από το 2010 στο 2019 έχει αλλάξει ο κόσμος μας. Το πρώτο μου ερώτημα λοιπόν είναι το εξή. Μήπως πρέπει να γίνει αναδιατύπωση της οδηγίας, γιατί έχει αλλάξει όλος ο κόσμος εδώ. Και ό,τι αφορά τις τεχνολογίες και ό,τι αφορά τις υπηρεσίες. Και τώρα αν έχουμε μια σειρά από εκτελεστικές πράξεις, ε, δεν είναι αυτή η κατάλληλη διαδικασία δεν εγγράφεται στα πλαίσια μιας ευρύτερης προσέγγισης. Ε, το δεύτερο σχόλιο μου τώρα. Με εκπλήσει και πάλι εδώ η διαδικασία. Θα μας ε, υποβάλλεται στις 13 Μαρτίου, είπατε, μια εκπληκτική πράξη ε, δύο εβδομάδες πριν κλείσει το κοινοβούλιο. Ε, αυτό με ενοχλεί με ενοχλεί πολύ από πλευρά διαδικασία. Δηλαδή, ε, έχουμε την εντύπωση εδώ ότι αυτό το μέτρο φτάνει σε μια στιγμή όπου το κοινοβούλιο εξαφανίζεται, έτσι. Και είναι πολύ έτσι, σοβαρή υπόθεση, ότι σοβαρό μέτρο. Αυτές οι συνεχόμενες πλαστικές πράξεις ε, για μια τέτοια οδηγία τη στιγμή ακριβώς που αλλάζει το κοινοβούλιο, τι να πω, Εμένα, εγώ έχω τι αμφιβολίε μου. Διότι, επαναλαμβάνω, θα έχει πολύ μεγάλες επιπτώσεις αυτή η απόφαση. Ε, συνήθως στις πράξει, πράξεις, καταξιδότητε πράξει, μιλάμε για, για τεχνολογική ουδετερότητα. Εσείς οι ίδιοι είπατε ότι δεν υπάρχει εδώ τεχνολογική ουδετερότητα. Ότι δεν τη σέβεστε. Ε, αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ εμένα. Ε, και με ενοχλεί, διότι αυτή η επιλογή είναι επιλογή με σημαντικό αντίκτυπο. Δεν λέμε απλά ότι θα μπορούσαμε να πάμε προς το Wi-Fi και ότι μετά αυτό θα οδηγήσει σε πρόοδο. Όχι, είναι μια επιλογή που θα δώσει έναν ολόκληρο προσανατολισμό, διότι δεν υπάρχει τη λειτουργικότητα με τις τεχνολογίες 5G. Αυτό δηλαδή που θα κάνετε εδώ δεν μπορείτε να το εφαρμόσετε αλλού. Γίνεται λοιπόν μια επιλογή συγκεκριμένη μια τεχνολογία ει βάρο μιας άλλης. Και αυτό με εκπλήσει διότι δεν είδα να υπάρχει κάποια μελέτη για το κόστος και για τον αντίκτυπο που θα είναι σημαντικά φαντάζομαι όλα αυτά. Και το κόστος της ανάπτυξης ε, και για τις υποδομές και για τις τεχνολογικές επιλογές Λέτε τώρα εσείς, ναι, αλλά αυτή η τεχνολογία, το ενδιαφέρον που παρουσιάζει είναι ότι είχε οριμάσει και μπορούμε να την αναπτύξουμε. Δεν βλέπω εγώ κάτι τέτοιο. Δεν βλέπω να έχει αναπτυχθεί, να έχει ε, επεκταθεί ως επιλογή ε, στα οχήματα. Και δεν μας το λένε αυτό ούτε τα κράτη-μέλη, ούτε ο κλάδος. Στην πραγματικότητα λοιπόν Εάν έχουμε έναν ανταγωνισμό μεταξύ των τεχνολογιών που είναι ότι, ότι η μία είναι όρημη και η άλλη δεν είναι, ε, δεν είναι ακριβώ έτσι τα πράγματα όπω τα παρουσιάζετε εσεί. Πόσο μάλλον ε, λέμε αν οι αποδόσει είναι οι ίδιε. Όχι, αν ακολουθήσουμε την επιλογή σα για το short range έχουμε WiFi, για το long range όμω θα πρέπει να ακολουθήσουμε ε, τεχνολογία 3G, 4G. Ε, έχουμε στην ύπαρξη δηλαδή, δύο λύσεων που διαφέρουν και σε επίπεδο υποδομών. Είναι αυτή η καλύτερη επιλογή ε, ανταγωνιστικά και παγκοσμίω. τίποτα, δεν μας εγγυάται αυτό. Η Κίνα δεν έκανε αυτή την επιλογή, έτσι. Να το λάβουμε υπόψη μας και αυτό. Και στις Ηνωμένε Πολιτείε, στις Ηνωμένες Πολιτείες έγινε μια παρεμφερή συζήτηση που μάλλον οδηγεί προς το 5G τελικά. Η λύση δηλαδή ε, με μια ενδιάμεση φάση ε, στο, με το Wi-Fi δεν, ε, εντάξει, δεν αποκλείστηκε αλλά χάνει έδαφος. Οπότε πολλά, πολλά είναι τα ερωτηματικά που δημιουργούνται στην υπόθεση αυτή. Και για το γεγονός ότι δεν υπάρχει τεχνολογική ουδετερότητα και γιατί η συζήτηση δεν είναι σαφής σε ό,τι αφορά τα συμφέροντα και των δε. Και το τελευταίο που θα πω και θα σταματήσω εδώ γιατί εντάξει θα είχα και άλλα να πω αλλά θα σταματήσω εδώ. Όλοι επιμένουν στην αναγκαιότητα ε, να θεσπίσουμε το 5G στην Ευρώπη. Φαίνεται να υπάρχει μάλιστα μια ε, ε, επιτάχυνση αυτής της διαδικασίας. Αυτή η επιλογή δεν αποθαρρύνει ε, την αναγκαιότητα της ε, ε, επέκταση του 5G. Φυσικά και το αποθαρρύνει. Ένα μέρος του πεδίου εφαρμογής εδώ εκεί οδηγεί. Εάν κάνω 5G μόνο για τα τηλέφωνα ή για τις τηλεπικοινωνίες, δεν είναι το ίδιο Εάν αυτή η εφαρμογή ε, είναι αναγκαιότητα ευρύτερη. Έτσι λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι εδώ υπάρχουν πολλοί λόγοι να το σκεφτούμε πολύ προσεκτικά το ζήτημα. Ε, είναι μια διαδικασία όπου ε, τα πράγματα γίνονται βεβιασμένα. Δεν συνηθίζουμε να το κάνουμε αυτό. Δεν συνηθίζει να το κάνει αυτό η Κομισιόν. Και υπ' αυτέ τι συνθήκε, βεβαίω, εντάξει, η συζήτηση συνεχίζεται, αλλά δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι έχει νόημα, ότι είναι σωστό να, να κάνουμε αυτή την επιλογή έτσι βεβαιασμένα. Ευχαριστώ κύριε Ρικέ. Είχα ζητήσει και εγώ να πάρω το λόγο εκ μέρους των Πρασίνων. Δεν θα επαναλάβω όλα όσα υπόθηκαν, αλλά ε, για τα διαδικαστικά εγώ δεν καταλαβαίνω την Κομισιόν γιατί δεν ήρθατε να μας δείτε και να μας πείτε όλα αυτά που μας είπατε πριν από ένα χρόνο. Αυτό είναι το πραγματικό ερώτημα. Γιατί εντάξει, καλά κάνουμε και το συζητάμε σήμερα, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι από άποψη ε, ρυθμιστική υπάρχει μια διαδικασία. Οπότε έχετε έρθει λίγο καθυστερημένα. Γιατί αυτή η καθυστέρηση. Διότι έχουμε τους δύο μήνες που προβλέπονται από την νομοθεσία για να ασκήσουμε το δικαίωμα εξέτασής μας για τις κατεξοδότητες πράξεις. Και εδώ τώρα ή πρέπει να δημιουργήσουμε μια εξαίρεση ή να τηρήσουμε τους κανόνες. Και ως πρόεδρος εγώ θα σας πω το ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε με το διαδικαστικό ζήτημα και γρήγορα μάλιστα. Το δεύτερο Συμφωνώ με τον κύριο Ρικέ. Είπε πολλά, αλλά έχει δίκιο επί της ουσίας και έθεσε ένα θέμα το οποίο πρέπει να θίξουμε. Λέτε στο έγγραφο που στείλατε την περασμένη Παρασκευή ότι η τεχνολογία της 5G ε, υπάρχει ήδη στην Ευρώπη. Αυτό γράφετε στον εγγραφό σας και θα ήθελα να μου πείτε Μπορείτε να μας πείτε σήμερα πού και από ποιον έχει εφαρμοστεί και ποια είναι τα αποτελέσματα. Και δεν θα πω κάτι άλλο. Κύριε Κόρ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Την τελευταία φορά που είχαμε συζητήσει στην Επιτροπή μας αυτό το ζήτημα, δυστυχώς δεν είχα ε, παρευρεθεί. Αλλά από ό,τι γνωρίζω, ε, συζητήθηκε και αναφέρθηκε πολύ συχνά αυτή η έννοια της ουδετερότητας τεχνολογικής. Όμως, ε, ε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι που χρησιμοποιήσατε αυτόν τον όρο, πρέπει να σας πω ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, η ουδετερότητα η τεχνολογική είναι πάρα πολύ σημαντική για μας που συμμετέχουμε στη χάραξη τη πολιτική. Αλλά ξέρετε τι άλλο είναι πολύ σημαντικό να μην επαρεμποδίζουμε την έναρξη ορισμένων project αναφερόμενοι απλώς ε, και μόνο ε, στις νέες τεχνολογίες και δίνοντας έμφαση σε αυτές. Ε, δηλαδή αυτό που χρειαζόμαστε είναι από τη μία πλευρά επικοινωνία ε, ή μάλλον ε, επικοινωνία από, τη, από την πλευρά των οχημάτων αφενός και ε, την υποδομή αφετέρου. Και νομίζω πως με τη σημερινή τεχνολογία έχουμε αυτή τη δυνατότητα να το κάνουμε γιατί ε, ήδη αξιοποιείται από ορισμένα οχήματα και είναι και εξαιρετικά σημαντική και για την αυτοματοποιημένη οδήγηση. Βέβαια δεν θα πρέπει να πούμε ότι ε, θα εστιάσουμε σε μία μόνο τεχνολογία, θα πρέπει να ορίσουμε πρότυπα με βάση ε, ε, την οποία θα υπάρχει και διαλειτουργικότητα και backward compatibility, δηλαδή συμβατότητα με προηγούμενε εκδόσει. Δηλαδή, οποιαδήποτε νέα γενιά τεχνολογία θα πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνεί με την προηγούμενη γενιά τεχνολογία. Δηλαδή, αυτό είναι και το ζητούμενο. Ένα δηλαδή σύστημα να μπορεί να επικοινωνήσει με ένα διαφορετικό σύστημα από άλλο όχημα το οποίο προέρχεται από άλλο κράτος μέλος. Δεν μας ωφελεί σε τίποτα μια τεχνολογία όταν αυτή είναι ενσωματωμένοι σε ορισμένα και μόνο νέα οχήματα, τα οποία όμω δεν είναι σε θέση να επικοινωνήσουν με άλλα οχήματα. Σε τίποτα δεν ωφελεί μια τέτοια τεχνολογία. Η ε, Επιτροπή ε, θεωρεί πω αυτά τα πρότυπα στην κατεξοδότηση πράξη θα ε, ωφελήσουν στην αύξηση τη οδική ασφάλεια. Ε, πραγματικά θεωρώ πως υπάρχουν 25.000 διαφορετικοί ε, λόγοι που μας κάνουν να επιμείνουμε σε αυτή την πρόταση της Επιτροπής και 25.000 είναι ακριβώς οι θάνατοι που έχουμε κάθε ε, χρόνο σε οδικά τυχήματα. Ευχαριστώ κύριε Τζαν Μίντερμπουργκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Κόχ. Διότι αν πάτε να δείτε το non-paper μιλάμε για το CITS από το 2016 τότε παρουσίασε τη στρατηγική της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε α μην προσποιούμαστε ότι δεν έχουμε ξαναδεί αυτό το θέμα και την πρώτη φορά που το βλέπουμε και ότι τώρα πρέπει να το διεκπαιρώσουμε στα γρήγορα. Ε, όπως μας λέει η Κομισιόν, εδώ και δύο μήνες ε, στην Επιτροπή αυτή έχουμε συζητήσει για αυτό το θέμα. Ε, χρειάζεται να καταλήξουμε κάπου και για τις επιχειρήσεις μας ώστε να μπορέσουν να κάνουν και τις απαραίτητες επενδύσεις. Το άρθρο 33 αυτής της κατεξουσιοδότησης πράξης λέει ότι η Κομισιόν θα μπορεί να καθορίσει νέες απαιτήσεις ε, για τις νέες τεχνολογίες. Με λίγα λόγια, αυτό που είναι σημαντικό είναι αυτή την τεχνολογική ουδετερότητα να μην την βάλουμε ως αντίπαλο αλλά να τη χρησιμοποιήσουμε για να έχουμε αποτελέσματα υπέρ των συμφερόντων των επιχειρήσεων γιατί όπως είπε και η Κομισιόν τίθεται θέμα ασφάλειας στο δρόμο, αποτελεσματικότητας ε, της ε, διαχείρισης της κυκλοφορίας, της οδικής κυκλοφορίας, μείωση των εκπομπών σωματιδίων και διοξιδίου του άνθρακα. Οπότε χρειαζόμαστε αυτά αποτελέσματα. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να μας βάζουν εμπόδια, να υπάρχουν εμπόδια αυτές της πράξης. Ε, αυτό δεν θα το δεχτώ. Μετατίθεται, υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα που έχει προβλεφθεί για την κατεξοδότηση ε, πράξη μέσα Μαρτίου, τέλη Μαρτίου που θα στέλνετε, θα σταλεί στο Κοινοβούλιο. Ελπίζω οι συνάδελφοι να μεριμνήσουν ώστε να τεθεί σε ισχύ η πράξη αυτή, ώστε να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί ω Ευρώπη και με τον υπόλοιπο κόσμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαν Μίλτεμπουργκ, Κύριε Ντεπρέ. Όχι, συγγνώμη. Ε, κύριε Βέργενεν, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ε, επιτρέψτε μου να πω και εγώ δύο λόγια σε ό,τι αφορά την τεχνολογική ουδετερότητα η οποία αναφέρθηκε επανειλημμένα, την ανέφερε και ο κ. Βαντεκάμπ και η Επιτροπή είπε ότι δεν είναι και απόλυτα ουδετερό. Οπότε σε κάθε περίπτωση η κατεξοδότηση πράξη μα θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με την Ευρωπαϊκή Στατική ITS και κατά συνέπεια θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα ε, ε, υβριδικό μείγμα τεχνολογιών ευθύ εξ αρχής η Επιτροπή μας είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι ε, τεχνολογικά ουδέτερη σχετική πράξη. Οπότε, αν ρίξουμε μια ματιά στην, στην σημερινή διατύπωση βλέπουμε ότι μόνο η ITS5 θεωρείται ως ε, συμβατή τεχνολογία, ενώ υπάρχουν πολλές ε, ε άλλες τεχνολογίες σε ITS. Υπάρχουν, για παράδειγμα, διαφορετικές τεχνολογίες οι οποίες χρησιμοποιούν ε, κινητή την τηλεφωνία, τα σχετικά δίκτυα, δηλαδή 3G και 4G. Οπότε νομίζω πως θα πρέπει να τηρήσουμε τη στάση που έχουμε ε, αναπτύξει, αν θέλετε, και έχουμε χαράξει με την ε, ε σχετική μας ε, στρατηγική, ότι δηλαδή ε, θέλουμε πλήρες υβριδικό μείγμα τεχνολογιών και τεχνολογική ουδετερότητα. Αλλά βέβαια άκουσα και τα διάφορα άλλα μέλη εδώ της Επιτροπής που έχουν διαφορετικές απόψεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ντεπρέ. Έχετε το λόγο για να απαντήσετε στο συνολό των ερωτημάτων σας. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, για την ε, οδηγία CITS. Α, κατά πόσο είναι ξεπερασμένη. Όχι, δεν είναι ξεπερασμένη σε καμιά περίπτωση. Πιστέψτε με. Ε, στα πλαίσια της οδηγίας CITS, στην αρχή έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο. Ποτέ δεν έχω δει μια νομοθεσία όμως τόσο ε, αθεκτική στις εξελίξεις. Ε, θέλω να επιμείνω εδώ εξετάσαμε θέμα ε, πρόσβαση δεδομένων πολύ νωρίτερα από άλλους. Έχουμε ένα πλήρες σύστημα τώρα για την, προστασία δεδομένων, για την ε, πρόσβαση δεδομένων στο πλαίσιο αυτό. Πολλές start-up, πολλοί πάροχοι πληροφοριών ε, ή πληροφορίες κυκλοφορία σε, σε πραγματικό χρόνο, ψηφιακοί χάρτες, αυτά χρησιμοποιούν αυτοί οι υπάρχοι χρησιμοποιούν αυτό το σύστημα, αυτή την, αυτό το, κανονισμό που υπάρχει από το 2010. Έτσι. Πρέπει να το πούμε αυτό. Ήταν από τις πιο καινοτόμες ε, πράξεις ε, ε, και πρωτοποριακές που έχω δει. Και ξέρω ότι το Κοινοβούλιο έκανε πολλά γι' αυτό. Εκεί βεβαίως που δεν ε, ήμασταν προνοητικοί ήταν οι κανόνες. Χάρη όμως το Κοινοβούλιο μπορέσαμε να το δούμε αυτό, να το δούμε, να το συνδυάσουμε και με άλλες, ε, άλλους τρόπους μεταφοράς. Αυτό που ήθελα να πω τώρα, ήθελα να επανέλθω στο εξή, διότι ακούω ε, ότι εδώ έχουμε ένα, μια μάχη μεταξύ 5G και του νέου αυτού συστήματος. Ε, θέλω να, μια στιγμή να ξαναδούμε το, το χάρτη, το γράφημα και να επανέλθω και σε αυτό που είπε ο κ. Βίρκανεν. Ε, δεν περιορίζουμε εμείς εδώ τίποτα. Δεν περιορίζουμε τη χρήση και τις λύσεις ε, Wi-Fi. Αντιθέτως, ε, πρέπει να εξηγήσω και γιατί γίνεται αυτό αυτή τη στιγμή, έτσι. Θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει αυτό σε μια άλλη στιγμή, χωρίς να λάβουμε όμως υπόψη μας τι θα μπορούσε να συμβεί στα διάφορα κράτη-μέλη. Για μια φορά προσπαθήσαμε να αναφερθούμε έξυπνα. Είπαμε Ας χρησιμοποιήσουμε την ε, δυνατότητα Connecting Europe, ας έχουμε διάφορα πιλωτικά προγράμματα σε διάφορα κράτη-μέλη. Αυτά τα πιλωτικά προγράμματα μεγάλωσαν με τον καιρό. Επτά κράτη-μέλη ε, ε, αναπτύσσουν λύσεις που χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνολογίες μόνο που σε αυτή τη φάση δεν ήμασταν σε θέση να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία εναρμόνισης για το 4G και το 5G. Η επόμενη μεταρρύθμιση της ε, πράξης εξουσιοδότησης θα καλύψει ακριβώ αυτό. Αυτό είναι βέβαιο. Μην έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Οι συνάδελφοι στα κράτη-μέλη εργάζονται προ την κατεύθυνση αυτή και με τον κλάδο. Όπω βλέπετε και στον πίνακά μα είναι κάτι που έχει προβλεφθεί ήδη. 5G τώρα και 5G2. Ακούστε με, και αυτό είναι μέρος μιας αφήγησης, έτσι. Πάμε πίσω στο σχέδιο δράση για το 5G. Ε, τότε ήδη υπήρχε συμπληρωματικότητα των διαφόρων τεχνολογιών. Επενδύουμε εκατομμύρια στο 5G. Γιατί, μόνο για την τεχνολογία. Θέλουμε κάποια στιγμή να μπορέσουμε αυτές τις νέες τεχνολογικέ εξελίξεις να τις ε, ε, ενσωματώσουμε και να έχουμε περισσότερες λύσεις στη διάθεσή μα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θέλουμε να συμβεί. Το συντομότερο δυνατόν μάλιστα. Ε, αυτό που θα είναι κάπως πιο δύσκολο είναι ότι εδώ έχουμε μια συσκευή που δεν έχει 5G και ζητώ από τις ε, συσκευές τις σημερινές να μου πούν τι θα συμβεί κάποια στιγμή αργότερα. Αν ήταν έτσι τα πράγματα θα είχαμε πολλούς πελάτες που ζητούν υπηρεσίες, ζητούν λύσεις που δεν υπάρχουν ακόμα. Λοιπόν, κατά πόσο θα πρέπει ε, να περιμένουμε ή αν είμαστε στο τέλος μιας διαδικασίας. Ίσως να ολοκληρώνεται η πρώτη φάση ε, στο τέλος αυτής της διαδικασίας. Ναι, ήταν όμως μια ε, ενδελεχής προσπάθεια. Τέσσερα χρόνια τώρα ασχολούμαστε με το θέμα αυτό. Πιστέψτε με. Και αντί να έρθουμε αμέσω με την πράσινη εξουσιακή προσπαθήσαμε όντως να δώσουμε μεγαλύτερη ε, ορατότητα σε ένα ευρωπαϊκό, σε ένα κείμενο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, μια ευρωπαϊκή στρατηγική στο τέλο του 2016. Και πήρατε θέση από αυτού του εγγράφου. Το συζητήσαμε. Συζητήσαμε τα ζητήματα αυτά σχετικά πρόσφατα. Κατά πόσο θα έχουμε τις ίδιες υπηρεσίες με το 4G. Ίσως όχι. Ίσως να έχουμε πιο προχωρημένες υπηρεσίες. Είναι πρόβλημα αυτό. Όχι, δεν είναι. Είναι πρόθεσή μας να το ενσωματώσουμε. Τώρα, η συμβατότητα εκ των υστέρων, αυτό είναι πρόβλημα, όντως. Αλλά αυτό δεν σημαίνει, και θέλω να το αναδιατυπώσω αυτό, αποφασίσαμε να μην περιμένουμε άλλο. Δεν λέμε ότι θα περιορίσουμε τον αυτό μας με μία μόνο τεχνολογία εδώ. Δεν πρέπει δηλαδή να το δείτε όσο ότι δεν λαμβάνουν υπόψη άλλες τεχνολογίες ή ότι διαλέγουμε ε, να φέρουμε στην παράθεση της ε, τεχνολογίας μεταξύ τους. Να προσθέσω κάτι εδώ. Δεν αντιμετωπίζουμε εμεί το φάσμα ε, με αυτό το κείμενο. Δεν είναι άλλωστε η εντολή μας. Εξετάζουμε πώς θα εξασφαλίσουμε την πρόσβαση στο φάσμα για το Urban Rail ε, δεν πρόκειται αυτό να ε, αλλάξει ή να ε, διαταραχθεί από, το, την νομοθετική πράξη αυτή. Κάτι άλλο τώρα, άρθρο 33. Να πω ότι εμείς είμαστε ανοιχτοί προς τις τεχνολογίες αυτές και έχουμε, εξοπλιζόμαστε πάση για να είμαστε όσο γίνεται πιο ανθεκτικοί να μπορούμε όσο γίνεται πιο γρήγορα να ενσωματώσουμε ε, καινούρια στοιχεία. Θα υπάρξει ανάλυση, θα υπάρξει συζήτηση. Αυτό έχει σχέση και με την ομάδα εμπειρογνωμόνων που μας ζητήσατε να είναι ανοιχτή αυτή η ομάδα και αυτό κάνουμε. Λοιπόν, πού λαμβάνει η χώρα αυτή η ανάπτυξη σε πολλά κράτη-μέλη. Σε πολλά κράτη-μέλη. Αυτό που λαμβανει η χωρα αυτη η αναπτυξη σε πολλα κρατη μελη σε πολλα κρατη μελη αυτο πρεπει να σας πω ίσως είναι ότι μέσω του μηχανισμού Connecting Europe έχουμε δώσει μεγάλη έμφαση στα κράτη-μέλη έτσι ώστε να λάβει η χώρα αυτή η ανάπτυξη εναρμονισμένα. Πολλές από τις δραστηριότητε μας λοιπόν και πολλές από τις τεχνικές προδιαγραφές που βλέπετε εδώ δεν είναι δικό μας αποτέλεσμα μόνο. Έχουν αναπτυχθεί με τη βοήθεια και την πραγματογνωμοσύνη και τις, ε, όσων τρέχουν τα προγράμματα. 16 κράτη-μέλη συμμετέχουν. Το λέω αυτό γιατί τη στιγμή που μιλάμε για εναρμόνιση, για εναρμονισμένους κανόνες, η ανάπτυξη θα είναι μαζική, θα είναι γρήγορη και μαζική. Πραγματικά υπάρχει μια πολύ σημαντική βάση πλέον για να προχωρήσουμε. Και τέλος, α ναι, ναι κυρία Ντεπρέ μπορείτε να μας πείτε γιατί ε, δεν σας αρέσουν, ε, ποια, είναι τα κρατη ναι η Γερμανία, να περάσω ξανά στα αγγλικά λέει κυρία Ντεπρέ, δεν ξέρουμε γιατί, δίνει το λόγο στον συνάδελφό της. North and South of Europe are part of ε, σε αυτή την πλατφόρμα συμμετέχουν ε, όλα τα, όλες οι χώρες δηλαδή της ε, Ανατολικής, της Βορρής και της, ε, Ευρώπης, οπότε έχουμε 65 συμπληρωματικές χώρες οι οποίες συμμετέχουν σε αυτή την πλατφόρμα. Το Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία, η Σλοβενία, η Αυστρία, η Ελβετία ως συνδεδεμένη χώρα, η Τσεχία, η Γερμανία, οι κάτω χώρες, το Βέλγιο, η Ουγγαρία, η Δανία, η Σουηδία, η Φιλανδία και μετά τη ε, Ζηλανδία ως συνδεδεμένη χώρα. Να μας πείτε καλύτερα εκείνοι που δεν, οι χώρες που δεν συμπεριλαμβάνονται. Θα ήταν πιο γρήγορο η απαριθμίση. Απάντηση. Ναι, ε, Πρόεδρε, υπάρχουν κάποιε χώρε τη Ανατολική Ευρώπη που προετοιμάζουν αυτή την περίοδο την προσχώρησή του στην πλατφόρμα. Και ένα τελευταίο σχόλιο σε ό,τι αφορά το non-paper σε σχέση με το ερώτημα που θέσατε. Σας στείλαμε το ταχύτερο δυνατό τις ε, ε, πληροφορίες ε, που περιλαμβάνονται εκεί, αλλά δεν περιλαμβάνονται εκεί οι πληροφορίες από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε ναι, θα, δείτε πότε θα είναι έτοιμη η πλέον νομοθετική πρόταση και εκεί θα περιλαμβάνονται τα πάντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Ντεπρέ. Όσον αφορά λοιπόν το χρονοδιάγραμμα, μας επιβεβαιώνεται ότι την κατεξουσιοδότηση πράξη θα την έχουμε στις 13 Μαρτίου. Είναι βέβαιο. Ωραία. Κυρία Μάισνερ, έχετε το λόγο, θέλετε να πείτε κάτι. Ναι, σα ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω και εγώ σύντομα να κάνω την παρέμβασή μου. Νομίζω πριν από 10 χρόνια κανένα δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι θα μπορούσαμε να συζητούμε μια τεχνολογία ε, ε, επικοινωνία μεταξύ των οχημάτων, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση τη οδική ασφάλεια. Όμω πραγματικά αυτή τη συζήτηση κάνουμε και σε ό,τι αφορά τη τεχνολογική ουδέτερα, ε, το είπα και προηγουμένω. Πάντοτε είμαι υπέρ τη τεχνολογική ουδέτερα, όταν υπάρχουν οι απαραίτητε τεχνολογίε. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την μείωση των εκπομπών άνθρακα, έχουμε το υδρογόνο, έχουμε όλε τι διαφορετικέ τεχνολογίε. Οπότε εκεί πράγματι χρειαζόμαστε τεχνολογική ιδιαιτερότητα. Αν όμω εδώ τώρα σε αυτό που συζητάμε έχουμε μόνο μία τεχνολογία, δεν μπορούμε να συζητούμε το ζήτημα τη τεχνολογική ιδιαιτερότητα αφού μόνο μία είναι διαθέσιμη τεχνολογία. Ξεκινάμε λοιπόν με αυτήν την τεχνολογία και από εκεί και μετά διασφαλίζουμε ότι στο μέλλον θα είναι δυνατόν να ενσωματωθεί και η τεχνολογία 5G. Και όπω είπα και προηγουμένω, αν λάβουμε υπόψη μα το πώ επιταχύνεται ο τεχνολογική τεχνολογικής ανάπτυξης, ε, τότε ε, πραγματικά ε, δεν είναι δυνατόν να λαμβάνουμε πάντοτε υπόψη σε τις τεχνολογίες. Τώρα, απευθυνόμενο στον συνάδελφο Ερτούκ, ναι, είπε ότι δεν θα ήθελε να υπάρξει μια μεικτή εικόνα στο μέλλον. Θα ήθελε δηλαδή όλα τα συστήματα να επικοινωνούν μεταξύ του ανά πάση στιγμή. Εντάξει, νομίζω ποτέ δεν θα φτάσουμε στην τέλεια κατάσταση. Δηλαδή, πάντοτε θα υπάρχει μια στέρηση ενδεχομένω σε κάποιε τεχνολογίε. Ε, εντάξει, ε, και υπάρχει και το σύντημα δηλαδή της διαβίβαση των σχετικών δεδομένων μεταξύ των οχημάτων. Δεν θα μπορεί, δηλαδή ε, θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό για τους χρήστες των οχημάτων να ε, υποχρεούνται να, να χρησιμοποιήσουν ένα συγκεκριμένο σύστημα. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν ε, καλό θα ήταν ναι να υπάρχουν πολλάπλέ τεχνολογίες ώστε να μπορέσουμε να βασιστούμε στη τεχνολογική ουδετερότητα αλλά έτσι όπως έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή ουσιαστικά δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιτροπή και είχαμε και τη δυνατότητα να κάνουμε τη σχετική συζήτηση και νομίζω πως με βάση αυτό τον όρο θα μπορέσουμε να προλάβουμε να περάσει αυτή η πρόταση μέσα στο διαθέσιμο χρονικό διάστημα. Ευχαριστώ κυρία Μάισνερ. Μια τελευταία ερώτηση από τον κύριο Βαντεκάμπα. Πολύ γρήγορα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πρέπει να προσέξουμε μην πούμε κάτι λάθος διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντα λέει ότι υποστηρίζει στεναρά τις νέες τεχνολογίες, ε, το λέει και σήμερα επί χάρτου για το 5G και εγώ έχω ρωτήσει το άρθρο 33 αρκεί ώστε να είναι σαφές για όλους πώς, ε, με ποια ταχύτητα και με ποιες μεθόδους και με ποιους συμπρογνώμονες ε, θα εισαχθεί η νέα τεχνολογία. Ακόμη δεν έχω λάβει απάντηση για αυτή την ερώτηση. Μπορείτε να απαντήσετε την ερώτηση, Κομισιόν. Το έχουμε ξαναπεί και το επαναλαμβάνω η Κομισιόν είναι επεπισμένη ότι η τεχνολογία 5G θα διδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο και την υποστηρίζουμε, αλλά δεν μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον. Αυτό μπορούμε να κάνουμε είναι να πούμε πότε θα είναι διαθέσιμη, αλλά μας είναι αδύνατον σήμερα να πούμε πώς θα χρησιμοποιηθεί και για ποιες υπηρεσίες. Όταν λοιπόν η ρήτρα αναθεώρησης της κατεξοδότησης πράξης ορίζει ότι είμαστε έτοιμοι να λάβουμε αρχεία ανθρώπων που θέλουν να κάνουν αλλαγέ στον κανονισμό, όταν λέει ότι η Κομισιόν θα αναλύσει αυτά τα αρχεία χωρί καθυστέρηση, αδικαιολόγητη, αυτό ακριβώ θα κάνουμε, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώ θα λάβουμε, ούτε πότε. Αλλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε και έχουμε κάνει είναι να πούμε ότι θα τα αναλύουμε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Το δεύτερο που είπαμε είναι ότι εντός δύο μηνών το πολύ θα υποβάλουμε το αρχείο αυτό σε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων που πράγματι έχουμε διευκρινίσει ότι θα αποτελείται από όλους τους σημαντικούς ενδιαφερομένους από το δημόσιο και το ε, ιδιωτικό τομέα για αυτό το θέμα. Θα ξεκινήσουμε σε αυτό το πλαίσιο μια συζήτηση και αυτό που κάναμε επιπλέον, ενώ δεν το έχετε δει ακόμα, είναι, θα προσπαθήσουμε να ορίσουμε μια προθεσμία για το ταχύτητα με την οποία αυτή η αρχική ανάλυση μπορεί να γίνει. Αυτό που δεν μπορούμε όμως να κάνουμε είναι σήμερα να συμπεράνουμε και να λάβουμε μια απόφαση, διότι δεν ξέρουμε για ποιο πράγμα θα πρέπει να αποφασίσουμε. Και τέλος, πρέπει να σας πω ότι υπάρχει και ένα νομικό επιχείρημα εδώ. Η Κομισιόν έχει το δικαίωμα πρωτοβουλίας. Δεν μπορούμε να προδικάζουμε τη δική μας απόφαση όταν δεν ξέρουμε τι θα αποφασίσουμε ακριβώ, επί ποιου πράγματο δηλαδή θα λάβουμε απόφαση. Οπότε τι δεσμευτήκαμε να κάνουμε, να είμαστε ανοιχτοί, να είμαστε όπω έχουμε πει ε, κατά επανάληψη, έτοιμοι για αυτή την τεχνολογία που πιστεύουμε ότι θα έρθει, θα έχει παίξει σημαντικό ρόλο και μόλι εμφανιστεί θα την εξετάσουμε χωρί αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Αυτό μπορούμε να υποσχεθούμε και ούτω και θα πράξουμε. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το χρόνο που διαθέσατε να έρθετε εδώ να μας παρουσιάσετε κάποιες αποφάσεις οι οποίες ε, έχριζαν διευκρινήσεων. Θα ζητήσω από το σύνολο των συναδέλφων να παραμείνουν στην αίθουσα και θα ξεκινήσουμε, θα συνεχίσουμε μάλλον ε, και κλεισμένο το θυρών όμως όσοι λοιπόν δεν έχουν το δικαίωμα να είναι εδώ στα πλαίσια της ε, χειρισμένων θυρών συνάντησης να αποχωρήσουν παρακαλώ.